Καλώ darf ich ήρθατε. ξαναρχίζουμε. Στα γερμανικά θα μιλώ εγώ, οπότε ε, βάλετε και ακουστικά. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ακούν. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα ωραίο θέμα. Έρασμο για όλου. Το πρόγραμμα τη Ένωση για την Παιδεία, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την Νεολαία και τον Αθλητισμό. Θα συζητήσουμε πρώτη φορά την πρόταση τη Κομισιόν εδώ για την εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμό την περίοδο 2014-2020. Εδώ μεταξύ όλοι μάθαμε με πόδινο τρόπο ότι η πρόταση των προηγουμένων προγραμμάτων τώρα θα μπουν σε ένα ευρύ πρόγραμμα το διαβίου μάθηση για το μετοκομμένιους, Εράσμους, Λεωνάρντο Νταβίντσι, Κρούντβιχ για τους επιμέρους τομείς κατάρτισης, το πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας στην, ε, ε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Εράσμους Μούντους, Τέμπους και τα διμερεί προγράμματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και βέβαια το πρόγραμμα για τους νέους και το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δραστηριότητες Ζαν Μονέ και ένα χωριστό κεφάλαιο που είναι για τον αθλητισμό. Ε, εγώ θα παρουσιάσω τις πρώτες μου σκέψεις για το πρόγραμμα και τη δομή του. Τον Ιούλιο ε, θα συνεδριάσουμε λεπτομερέστερα και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα θα μιλήσουμε για διαχειριστικά και τεχνικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά στην πρόταση αυτή και μετά θα υποβάλω το Σεπτέμβρη την πρόταση ε, έκθεσης και αρχές Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. Όπως ξέρουμε όλοι δεν ξέρουμε πόσα χρήματα θα πάρουμε ακόμη, οπότε ό,τι κάνουμε θα παρουσιάζεται σε ποσοστά και μετά θα δούμε αρχές του χρόνου πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Καλώς. Το πρόγραμμα για το Lifelong Learning είναι καινούριο πολυετές πρόγραμμα, 7 ετών, θα το συζητήσουμε. Αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της στρατηγικής 2020 και των πρωτοβουλειών των εμβληματικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας από τους πέντε βασικούς στόχους στρατηγική 2020 είναι να μειωθεί σε λιγότερο από 10% το ποσοστό αυτών που διακόπτουν το, την εκπαίδευση και αυτών που ολοκληρώνουν και την τριτοβάθμια ή η ανώτερη η ανώτατη εκπαίδευση και ε, αυτό να αυξηθεί κατά 14% τουλάχιστον. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Κομισιόν έχει τώρα προβλέψει περισσότερα κονδύλια στον προϋπολογισμό ε, μεγαλύτερο ποσοστό, όταν είναι πολύ μικρό το ποσοστό βέβαια, α, δεν είναι πολύ, αλλά είναι 70% παραπάνω τα κονδύλια που προβλέπει η Κομισιόν. Εμείς συμφωνούμε και ελπίζουμε ότι τουλάχιστον στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό να είναι σαφές ότι χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το τίποτα αν πάει στο 70% αυτό είναι το αναγκαίο. Αν συγκρίνουμε τώρα τα άλλα προγράμματα, κοινωνικά ταμεία κλπ, ε, βλέπουμε πόσο μικροσκοπικό είναι το δικό μας ποσοστό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μείνει τόσο μικρό. Επειδή έχουμε υψηλούς στόχους στον τομέα, πρέπει να είναι και ψηλότερο το ποσοστό. Τώρα, οι μεγαλύτερες διαφορές και αλλαγές στο διαβίου μάθηση είναι ότι οι νέες ε, ε, πρωτοβουλίες συνοψίζονται στη νεότητα, εκπαίδευση ε, ΑΕΗ, Κομένιους Εράσμους, Λεοβονάρντο Νταβίντσι, εκπαίδευση ενηλίκων και Εράσμους Μούντους, Τέμπους και περαιτέρω διμερεί προγράμματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών. Και προστίθεται, όπως είπαμε, το πρόγραμμα Youth in Action. Επίσης έχουμε και τις δραστηριότητες Jean Monnet, χωριστό κεφάλαιο. Μια άλλη μεγάλη διαφορά είναι η αρχιτεκτονική της πρότασης Κομισιόν. Η Κομισιόν ήθελε να βρει μια ισορροπία μεταξύ εναρμόνισης και ευελιξίας Ήθελε και δραστηριότητες αλλά και τη διαχείριση του προγράμματος να την εξορθολογήσει και να την απλουστεύσει. Έτσι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει. Τώρα έχουμε τρεις τύπους δράσεων στο πρόγραμμα. Πρώτον, ε, κινητικότητα μεμονωμένων προσώπων. Δεύτερον, συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και των καταξιωμένων διαδικασιών. Και τρίτον, υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων η απλουστευσή, απλοποίηση είναι πρόσδεκτη Αυτό το θέλουμε πολύ ιδιαίτερα κατά, την, ε, κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων. Όμως οι συγκεκριμένες δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας δύσκολα μπορούν να ε, εντοπιστούν ιδιαίτερα ε, στο το κομμάτι για την νεολαία δεν, έχει, δεν είναι ορατό στη συνολική πρόταση. Η πρόταση προγράμματος για το, την νεολαία δεν έχει άρθρο ούτε δική της ενότητα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον θα υπάρχει προώθηση η οποία θα σκοπεύει στους επιμέρους στόχους, μέσα και δομές της ευρωπαϊκής εργασίας για τους νέους. Αν δεν υπάρχει κεφάλαιο χωριστό όχι, αν μπορεί να μην υπάρχει πρόγραμμα χωριστό. Χρειάζεται όμως η νεολαία δικό της κεφάλαιο στο πρόγραμμα και σαφή ξεχωριστό δικό της προϋπολογισμό. Και πρέπει να λέει ακριβώς ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα προαχθούν αυτονοήτως είναι σημαντικό ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν ικανότητες και ε, δεξιότητες σημαντικές για την αγορά εργασίας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτό. Δεν πρόκειται μόνο για την αγορά εργασίας. Πρόκειται και για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, για πολιτιστικά θέματα και για συμμετοχή στην κοινωνία που θα πρέπει όλα αυτά να τα προωθήσουμε και να τα αναφέρομαι επακριβώς στο πρόγραμμα. Δεύτερο σημείο, ο τίτλος Εράσμους, Εράσμους για όλους. Ο τίτλος δεν είναι κατάλληλος. Το Εράσμους είναι συνδεδεμένος με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κινητικότητα των φοιτητών. Και το όνομα είναι μια, ε, ένα ακρόνιμο. Σημαίνει European Action Scheme for the Mobility of University Students. Αυτό είναι το Εράσμους. Αυτό που είχαμε ως πρόγραμμα διαβίου μάθησης, αυτό που γνωρίζαμε ως διαβίου μάθηση, πάει πολύ πέρα από το πρόγραμμα Εράσμους. Για, στη διαβίου μάθηση ανήκει και η σχολική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση ενηλίκων και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι συνδεδεμένα με την κινητικότητα πάντα, ούτε μπορεί ούτε πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την κινητικότητα. Συνδέονται όμως με την περιφερειακή συνεργασία σχολείων στα πλαίσια του Κομένιου Ρέγγιο που είχε μεγάλη επιτυχία το, το τελευταίο πρόγραμμα. Εταιρικέ σχέσει, συμπράξει στην εκπαίδευση ενηλίκων και άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό ο τίτλο του προγράμματο δεν πρέπει να είναι περιοριστικό. Ακόμα κι αν ακούγεται ωραίο, περιλαμβάνει πράγματα που δεν μπορεί να τηρήσει. Το έρασμο για όλου, όταν ε, αναφέρεται ε, σε φοιτητέ είναι λάθος. Δεν υπάρχει έρασμος για όλους. Το εράσμος παραμένει ένα πρόγραμμα για εκείνους που έχουν τα χρήματα να συμμετέχουν. Παρακαλώ θερμά λοιπόν να το ξανασκεφτείτε μήπως το lifelong learning ε, θα έχουμε ένα καλύτερο ε, όνομα. Η Κομισιόν όταν πριν από 5-6 χρόνια δημιούργησε το πρόγραμμα αυτό, τότε ήταν lifelong learning. Δεν το εφεύραμε εμείς, η Κομισιόν το εφεύρε και μας άρεσε γιατί τα κάλυπτε όλα στον τομέα αυτών. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν πριν από 4-5 χρόνια. Γιατί αυτό που θέλει να κάνει τώρα είναι να συνδυάσει τους επιμέρους τομείς, να τους συγκεράσει. Και αυτό θα μπορούσε να το είχε κάνει και πριν από 4-5 χρόνια στα πλαίσια του lifelong learning. Άλλωστε, όταν είχαμε δώσει την έγκρισή μας, κάτι τέτοιο είχαμε υπόψη μας. Ε, πάμε τώρα στα ονόματα των, ε, της, της, του κάθε ε, επιμέρους προγράμματος. Θα πρέπει το όνομα να προωθεί την ταυτότητα. Γι' αυτό είναι σημαντικό το όνομα. Κομένιους για τη σχολική εκπαίδευση του Εράσμους, για την ε, τριτοβάθμια, Λεωνάρντο Νταβίντσι, ε, και Γκρούνβιχ για την ε, εκπαίδευση, ε, επαγγελματική κατάρτιση και ενηλίκων. Στους τομείς εκπαίδευσης που κάθε φορά αναφέρονται εδώ υπάρχουν ισχυρότατα δίκτυα τα οποία αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι δίκτυα χρηστών και οργανωτών που εδώ και χρόνια ασχολούνται και γνωρίζουν καλά τα προγράμματα αυτά. Πολλοί δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα Κομένιους, το ξέρω, το Εράσμους το ξέρουν όλοι. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν το Κομένιους. Το Κομένιους όμως δεν απευθύνεται σε μεμονωμένους μαθητές, αλλά σε σχολεία και δίκτυα που διευκολύνουν να λειτουργήσει το πρόγραμμα Κομένιους σε αντίθεση με το Εράσμους. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ θερμά να σκεφτείτε ότι όλα αυτά σε σχέση με τις επιθυμίες της και τις επιδιώξεις της Κομισιόν, ότι δηλαδή θέλει κάποιες διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους ε, προγραμμάτων, να μείνουμε εκεί. Και τα καταξιωμένα ονόματα, παρόλο που δεν είναι οικία σε μερικούς γιατί δεν δουλεύουν σε αυτό το τομέα, να τα διατηρήσουμε παρόλα αυτά. Πρόκειται για δραστηριότητες για τις δραστηριότητες που θα προωθηθούν μέσα από το πρόγραμμα συζητούμε ακόμη και πρέπει να συζητήσουμε πολύ. Η πρόταση της Κομισιόν παραμένει πολύ γενική, οπότε δεν είναι σαφές ποιες δραστηριότητες συγκεκριμένα θα προωθηθούν και ποιες όχι. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα και περισσότερες πληροφορίες, ούτως ώστε οι χρήστες του προγράμματος να αντικατοπτρίζονται στο νομοθετικό κείμενο. Την τελευταία φορά μου είπαν, να μέσα είναι, περιλαμβάνονται όλα. Εγώ όμως δεν τους βρήκα. Δεν είμαι εγώ πρόσκοπος που θα πάει να ψάξει στα μονοπάτια. Θέλω με μια ματιά να βλέπω τι είναι δυνατόν να, τι είναι δυνατόν να γίνει για αυτούς που ε, χρειάζονται το κομμένιος ε, και όλα τα άλλα. Θα πρέπει να γίνει πιο φιλικό προς τον χρήστη, με μεγαλύτερη ορατότητα και να, πιο εύκολα να βρίσκει κανείς αυτό που θέλει. Τώρα, για τη δομή της έκθεσης. Προτείνω να τροποποιήσουμε την πρόταση της Κομισιόν με την έκθεσή μας έτσι ώστε η εκπαίδευση, η κατάρτιση και αθλητισμός να χωρίζονται μεταξύ τους. Αυτό συγκεκριμένα θα σήμαινε ότι για κάθε τομέα θα υπάρχει χωριστό κεφάλαιο. Γενικά, γενική επαγγελματική εκπαίδευση είναι το ένα, η νεολαία είναι το δεύτερο, ο αθλητισμός θα είναι το τρίτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο γενική και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει τους διάφορους τομείς προγραμμάτων για την εκπαίδευση και να αναφέρει και τους επιμέρους ε, στόχους αυτών των προγραμμάτων. Η αρχιτεκτονική της πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει ως ένα βαθμό να διατηρηθεί, ούτως ώστε τα επιμέρους κεφάλαια να συνεχίσουν να κινούνται γύρω από τις δράσεις που προτείνει η Κομισιόν, δηλαδή κινητικότητα των επιμέρους προσώπων, η συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και των καταξιωμένων διαδικασιών και η υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό θα πρέπει να ε, αντικατοπτρίζει τη δομή αυτή. Όμως οι δράσεις 1 και 2 θα πρέπει για κάθε τομέα της εκπαίδευσης να περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες ποιες δραστηριότητες είναι αυτές που θα υποστηριχθούν. Παραδείγματα. Η δράση κινητικότητα μάθησης των επιμέρους προσώπων θα πρέπει να αναφέρει ότι με τον Εράσμου στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η κινητικότητα μεμονωμένων φοιτητών προωθείται για τις σπουδές και τις πρακτικές ασκήσεις ε, όπως και η κινητικότητα των ε, διδασκόντων ε, η συνεργασία για την πρόθεση της καινοτομίας και καταξιωμένων διαδικασιών θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, στο Κομένιους για παράδειγμα, θα δημιουργούνται συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ σχολείων για κοινά προγράμματα με στη συμμετοχή μαθητών και διδασκάλων. Η ε, περιφερειακές συμπράξεις που είναι γνωστές ως Κομένιους Ρέγγιο στον τομέα της ε, εκπαίδευσης ε, ενηλίκων. Κυρίως έχουμε εδώ πολυμερή προγράμματα και δίκτυα για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταλλαγής καταξιωμένων πρακτικών. Για τις δράσεις 1 και 2, δηλαδή κινητικότητα μάθησης και συνεργασία, τέτοιες λεπτομερείς περιγραφές θα πρέπει να γίνονται σε όλους τους τομείς. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις περιγραφές αυτές. Δύσκολο το έργο, αλλά οι συνεργάτες μας είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό. Πάμε τώρα στον τομέα νεολαία. Εδώ η αρχιτεκτονική της πρότασης πρέπει να είναι η ίδια. Με τρεις δράσεις. Πρώτον, κινητικότητα ε, μάθησης όλων. Ε, Επίση πάλι το ίδιο εδώ οι καινοτομίε και οι καταξιωμένε ε, πρακτικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Και στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι δραστηριότητες 1 και 2, δηλαδή ανταλλαγή νέων και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντική. Όλο το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να προσανατολίζεται στις ιδιαιτερότητες των αναγκών των νέων. Πάμε τώρα στον αθλητισμό. Υπάρχει ένα χωριστό κεφάλαιο για τον αθλητισμό. Αν το συγκρίνουμε με τα άλλα κεφάλαια βέβαια είναι ένα μίνι κεφάλαιο, μικρούλι. Αλλά αφού δεν έχει πολλά, πώς να βάλουμε εμείς. Εδώ οι χρήστες θα πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο μαζικό αθλητισμό grassroots, στη βάση. Η πρόταση αναφέρει, δεν αφαίρει όμως τον μαζικό αθλητισμό εξπρέσεις βέρμπης, πρέπει όμως, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η πρόταση επίσης ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό και τη συμβατότητα αθλητισμού και να προωθεί τη συμβατότητα αθλητισμού και εκπαίδευση. Μία από τι πέντε δραστηριότητε είναι η υποστήριξη μη εμπορικών αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να είναι δυνατή αν οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σαφή σχέση με τους στόχους που αναφέρονται στον τομέα, όπως προώθηση της, της κοινωνικής ένταξης ε, ε, μειονεκτικών ομάδων, παραολυμπιακή, ειδική ολυμπιακή και άλλα. Πάμε τώρα στις δραστηριότητες Ζαν Μονέ. Συνολικά έξι θεσμοί υποστηρίζονται εδώ για τις δραστηριότητες Ζαν ναι. Θα εξακολουθούν τα Jean Monnet αλλά στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Jean Monnet υπάρχουν έξι ε, ιδρύματα που θα προωθηθούν. Η Κομισιόν τα τέσσερα τα έβαλε στις ελληνικές καλένδες και κράτησε την ε, Μπρούζ και τη Φλωρεντία. Στο Μάστριχτε το Management Institute δεν υπάρχει, η Ακαδημία Δικαίου στην Trier δεν είναι, η European Agency for Development ε, Special Needs δεν είναι πια μέσα, ούτε το International Center of European Training στην Νίκαια. Αυτά βγήκαν απ' έξω. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως τα ιδρύματα αυτά όλα χρειάζονται διαρκή υποστήριξη. Δεν υπάρχει λόγος γιατί να κάνουμε διάκριση μεταξύ των πρώτων δύο και των υπολείπων τεσσάρων. Μου είπαν ότι αυτό γίνεται διότι στους άλλους τομείς στην αγορά υπάρχουν πολλοί και μεγάλοι ανταγωνιστές και δεν μπορούμε γι' αυτό το λόγο εμείς να υποστηρίζουμε συγκεκριμένα ιδρύματα αν ε, τραβάει και ισχύει για το, επιχείρημα αυτό της αγοράς, ισχύει και για την Μπρούζ και τη Φλωρεντία. Αυτά που διδάσκονται εκεί, ας πάρουμε την Μπρούζ. Εγώ την Μπρούζ την αγαπώ. Δεν θέλω να στερηθεί την υποστήριξη, αλλά αν ισχύει το επιχείρημα της αγοράς, το ε, Πανεπιστήμιο του Ζαρμπρούκεν είναι το ίδιο παλιό όπως της Μπρούζ και κάνει την ίδια δουλειά, καλή δουλειά και δεν πήρε ποτέ ούτε ένα σέντ από εμά. Ε, από τη σκοπιά του ανταγωνισμού λοιπόν καταρρύπτεται το επιχείρημα. Κάποια φορά είπα ή όλοι ή κανείς. Όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να πάρουν μια επιχορήγηση με προγράμματα, ε, με πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ε, όλοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν για να είμαστε δίκαιοι. Εν τω μεταξύ κάτι άκουσα ότι προς τα εκεί αποφάσισε και το Συμβούλιο. Είπε το Συμβούλιο όλοι να μετέχουν. Πάω τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ελάχιστα ποσοστά χρηματοδότηση για του επιμέρους τομεί. Ελάχιστα ποσοστά για τους στόχου εκπαίδευση, μόνο στη συνοδευτική ανακοίνωση περιλαμβάνονται, όχι στην πρόταση του κειμένου. Η... η ανακοίνωση δεν έχει όμως δεσμευτική ισχύ, άρα τα ελάχιστα ποσοστά θα πρέπει να περάσουν στο διατακτικό το ύψος αυτών των ελαχίστων ποσοστών πρέπει να τα συζητήσουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε. Στο πρόγραμμα Lifelong Learning αυτά τα ποσοστά μέχρι τώρα ήταν 82%. Και έχουμε και το Youth in Action συμπληρωματικά, επιπροσθέτως. Τώρα κάνουμε τους λογαριασμούς και η Κομισιόν προβλέπει μόνο 56% να τα κατανείμει στους τομείς. Η ανακοίνωση λέει για να διασφαλίσουμε ότι για τους σημαντικότερους ε, εμπλεκόμενους και παραλήπτες ε, θα διατίθενται τα ίδια κονδύλια όπως την περίοδο 2007-2013. Τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά προβλέπονται για τα προγράμματα στην εκπαίδευση ε, που δεν πρέπει να διαφοροποιηθούν προς τα κάτω, 25% για την εκπαίδευση, επαγγελματική και ανηλίκων 17%, 17% από αυτό είναι για τους ανηλίκους, α, όχι, και ανηλίκων 2%, σχολική εκπαίδευση 7%, νέοι 7%. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι το 90% πρέπει να επιμεριστεί. Εμείς έχουμε εκλεγεί ως πολιτικοί ε, εκπρόσωποι και θα πρέπει να καθορίσουμε τι θα γίνουν τα χρήματα αυτά, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Και δεν θέλω να έχω να πω κάτι για τα 56% όταν αναφέρεται στο, στο κείμενο και ε, για το 44% να αποφασίζουν οι αξιοσέβαστοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικοί. Αλλά τα χρήματα πώς θα τα δαπανούμε, θέλουμε να έχουμε και εμείς ένα λόγο. Έτσι είναι το Κοινοβούλιο, γι' αυτό μεταξύ άλλων εκλέγεται. Δεν εκλέγεται για να εξουσιοδοτεί ένα μη εκλεγμένο όργανο που κάνει καλή δουλειά και θα διαχειριστεί καλά τα, τα κονδύλια, αλλά δεν μπορεί να του δίνει αυτού του φορέα ε, εν λευκό επιταγή. Οι, εθνικές, οι εθνικοί οργανισμοί στο πρόγραμμα λέει ότι ένας οργανισμός σε μία χώρα θα είναι υπεύθυνο για όλα αυτά που συζητήσαμε. Νομίζω ότι ε, θα τα αφήσουμε λόγω της αρχής της επικουρικότητας στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν επιτόπου, είναι σαφές ότι μια χώρα δεν μπορεί να δαπανά για τη διοίκηση πιο πολλά από τα προβλεπόμενα. Μια χώρα όπως η Γερμανία που έχει οργανισμό για κάθε πρόγραμμα δεν έχω δει να έχει δώσει ούτε ένα σεντ παραπάνω. Ναι, εμείς έχουμε ένα γραφείο, όχι οργανισμό, ε, ένα γραφείο τους τομείς όπου εργαζόμεθα και σε εθνικό επίπεδο. Για το Εράσμους είναι οι ίδιοι άνθρωποι που επισκέπτονται και την ε, Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Υπηρεσία. Μέχρι τώρα ε, είδαμε ότι και το Συμβούλιο αποφάσισε από τον οργανισμό να κάνει οργανισμούς και ο καθένας έχει την ευχέρεια να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο σε επίπεδο κράτους μέλους. Είναι πολλά τα ανοιχτά ακόμα θέματα. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα, η Κομισιόν πρότεινε αύξηση 70 περίπου της 100 σε σχέση με το παρόν, δηλαδή 17,3 δις ευρώ συνολικά. Αυτό βεβαίω είναι ευπρόσδεκτο και με όλη μας την καρδιά το καλωσορίζουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε μέχρι την τελεσίδικη απόφαση για τον προϋπολογισμό όταν τελειώσουν οι διαπραγματεύσει για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Ελπίζω να τελειώσουν πριν από το τέλος του χρόνου, σε αντίθεση με το παρελθόν, για να τρέξει το πρόγραμμα για το 2014. Αν όμω πάνε στα μέσα ή στο τέλος της επομένης χρονιάς, τότε θα είναι δύσκολο να αρχίσει το πρόγραμμα να λειτουργεί το 2014. Common sense, κοινή λογική, ελπίζω να επικρατήσει και τα χρήματα που προτίθενται να δώσουν να τα δώσουν. Βέβαια είναι πολύ μικρό ε, το ποσοστό, είναι λίγα τα χρήματα, γι' αυτό ας φροντίσουμε μαζί με την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών και το Συμβούλιο, ας φροντίσουμε τα χρήματα που δαπανώνται να δοθούν. Γιατί το 70% σε σχέση με αυτά που είχαμε είναι πραγματικά ψίχουλα. Όλα ήταν, πήγαιναν στα διορθωτικά ταμεία, την ΚΑΠ κλπ. Ε, ένα άλλο πρόβλημα είναι το εξής. Όπως συζητήσαμε και μεταξύ μας και η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες προβλέψεις, στην αρχή είχα ενθουσιαστεί από τις προβλέψεις της Κομισιόν, αλλά μετά προσγειώθηκα λίγο. Ε, τώρα, είναι αυτό το Master Mobility Scheme. Να κάνει κανείς το Master του σε άλλη χώρα. Ολόκληρο το Master σε μια άλλη χώρα. Θα πρέπει να δοθούν πιστώσεις που θα τις δώσει η Τράπεζα Επενδύσεων. Και εμεί, στο πρόγραμμά μα θα δημιουργήσουμε γι' αυτό ένα ε, ταμείο εγγύησεων. περίπου 181 εκατομμύρια ευρώ θα ε, ενταχθούν εκεί στην αρχή, λιγότερα. Αλλά καθώς οριμάζουν οι πιθανές εγγύησεις, όπου δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε εμείς εγγύηση, θα πάμε στα 180 ε, εκατομμύρια ετησίως. Αυτά τα χρήματα δεν διατίθενται έτσι γενικώ, γιατί είναι ταμείο εγγύηση για εκείνου που δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν, γιατί μετά τι σπουδέ του δεν θα έχουν βρει ακόμη δουλειά. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό του προγράμματο. Πρόκειται για το 5% του προπολογισμού του προγράμματο. Αυτά ήταν οι γενικέ παρατηρήσει από μένα. Αυτό είναι ο προβληματισμός μου Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, αλλά ήθελα γενικά να περιγράψω το πρόγραμμα, πώς το βρίσκω, ε, καλές προσεγγίσεις έχει, ε, ορισμένες φορές ε, βλέπω ότι χρειάζεται βελτιώσεις όπως σας είπα και για τα επιμέρους, όπως δηλαδή τι ακόμη είναι σημαντικό στα πλαίσια του Εράσμους, όπως η πρόθεση της Θερινής Ακαδημίας ή ότι θα πρέπει οι υποτροφίες να μην δίνονται για λίγους μήνες, αλλά στα πλαίσια της κινητικότητας του Εράσμους να δίνονται για ένα ή δύο χρόνια. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που θα τα συζητήσουμε από τον Ιούλιο και από τον Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε κατατεθειμένο μπροστά μας το πρόγραμμα. Τότε θα κάνουμε τροπολογίες και θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Τώρα, δεν θα κάνουμε προσπάθειες να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά τη γενικότερη δομή που υπάρχει νομίζω και στα αγγλικά. Ας κάνουμε μια συζήτηση, έχουμε μισή ώρα καιρό και μετά θα κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ έπρεπε να σας τα πω όλα, αλλά νομίζω ότι έκανα γρήγορα. Δεν θα επαναλάβετε αυτά που είπα, μόνο στα σημεία που έχετε κριτική θα παρέμβετε και αυτά θα πείτε. Η... Σκιώδης. Ναβιντάλοβα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε η συγκητριά μας και πρόεδρος. Και εμείς θα θέλαμε να το είχαμε συζητήσει νωρίτερα. Ήδη κάναμε μια συνάντηση και συμφωνήσαμε για κάποια πράγματα. Όπως είπατε και χαίρομαι που το θίξατε, υπάρχουν αυτοί οι τρεις στόχοι, οι τρεις τομείς νεολαία, αθλητισμός και εκπαίδευση. Ήμουν πολύ απογοητευμένη με την αρχική σας πρόταση, όπου η νεολαία είχε βγει από την πρόταση της Κομισιόν, τουλάχιστον δεν φαινόταν αρκετά. Χαίρομαι λοιπόν που οι βασικές αρχές, οι βασικοί άξονε τώρα είναι πιο ξεκάθαροι. Το πρόγραμμα για την νεολαία και η νεολαία είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που επιτέλους συμφωνήσαμε γι' αυτό. Για τα ελάχιστα, 90%. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει η Κομισιόν για το μισό απ' όλα. Εμείς θέλουμε να αποφασίσουμε το μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού. Και ελπίζουμε να δούμε τις αυξήσεις που θα μας ικανοποιήσουν. Η απασχόληση ήταν ένας από τους στόχους της Κομισιόν ή μάλλον καλύτερα η απασχολησιμότητα. Όταν μιλάμε για την εκπαίδευση, την νεολαία και την, τον αθλητισμό, δεν είναι μόνο η απασχολησιμότητα που είναι σημαντική. Υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι σημαντικά. Το έρασμος για όλους είχε και άλλους στόχους. Η εκπαίδευση Δεν είναι μόνο να πάρει κανεί ε, στα 30 του ένα πτυχίο πανεπιστημίου και να μην το κάνει τίποτα. Η διαβίου μάθησε είναι ακριβώ αυτό που λέει ο όρο. Μαθαίνω συνέχεια όσο ζω, ανεξάρτητα από την ηλικία μου και από το θέμα. Και επομένω θα πρέπει να δοθούν κονδύλια. Οριζόντια σε όλε τι κοινωνικέ ομάδε. Δεν μπορούμε να έχουμε την κατάσταση όπω το Εράσμου, όπου μόνο μια ελίτ, μόνο η πλούσια ελίτ ε, εποφελείται από τις επιχορηγήσεις και από την οικονομική υποστήριξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η νεολαία είναι πολύ σημαντικό και οι οργανώσεις των νέων. Στο Erasmus for υπάρχουν τα επιχειρησιακά κονδύλια, επιχειρησιακές επιχορηγήσεις. Και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Δεν μιλάω μόνο για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την νεολαία εδώ. Αν αυτές οι επιχρησιακές επιχορηγήσεις ε, ε, εξαφανιστούν, τότε θα εξαφανιστούν και οι οργανώσεις νέων. Γιατί δεν θα έχουν λεφτά πια να συνεχίσουν να λειτουργούν. Σε πολλά συμφωνώ μαζί σας. Για τις εθνικές ε, συντονιστικές υπηρεσίες θα πρέπει να κρατήσουμε το status quo. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε νέες δομές, να επανεφεύρουμε πράγματα που υπάρχουν. Μια και έχουμε, όταν έχουμε δομές που λειτουργούν, ας τις ε, διατηρήσουμε, ας κρατήσουμε τα παλιά που λειτουργούν. Ευχαριστώ κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ Ντόρις, ευχαριστούμε για την εκτενέστατη και σαφή παρουσίαση την αξιολόγηση των προτάσεων, την κριτική. Να πω και εγώ δύο λόγια. Χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η δημοσιονομική αύξηση του 70% και τώρα στην κρίση και την ανεργία των νέων ε, στα κράτη-μέλη είναι σωστή πολιτική προσέγγιση το πρόγραμμα αυτό και στον τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης ε, στα προγράμματα νέων πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Να πω όμως ότι οι 8 payer ε, κράτη-μέλη ζητούν στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο περικοπή κατά 10%. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση αυτή δεν είναι καθόλου σίγουρη. Θα ε, γίνουν σκληρές αντιπαραθέσεις. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε το παν να περάσει η πρόταση αυτή. Όλα τα άλλα είναι μια μειοπική και λανθασμένη πολιτική. Αλλά δυστυχώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις απειλές που υπάρχουν και ότι μπορεί ενδεχομένως τα νούμερα να είναι διαφορετικά. Μικρότερα δηλαδή, ελπίζω να τα αποφύγουμε. Τόνισες επίσης ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, αλλά μπαίνει και θέμα προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης, μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί αυτή είναι και η ανθρωπιστική παιδεία η οποία στοχεύει στη βελτίωση όλων. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε πάντα στα προγράμματα. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν απεικονίζει όλες αυτές τις συνιστώσεις. Τώρα για τον τίτλο. Με το Εράσμους για, Εράσμους για όλους η Κομισιόν υποθέτει ότι είναι σωστό γιατί το Εράσμους ήταν μια επιτυχία και θέλει να συνεχίσει να το ε, προωθεί. Είναι δημοφιλές. Αναμφίβολα είναι επιτυχημένο το Erasmus πρόγραμμα, αλλά είναι λάθος να ονομάσουμε όλο το πρόγραμμα έτσι, διότι δεν πρόκειται για το Erasmus for All, δεν είναι κάτι τέτοιο το πρόγραμμα αυτό και επίσης άλλα πολύ σημαντικά προγράμματα δεν θα είναι πια τόσο ορατά αν επιλέξουμε αυτή τη γενική ονομασία υπάρχουν λοιπόν, ή, θα πρέπει να γυρίσουμε στο παλιό όνομα, lifelong learning, για να ξέρουμε ποια προγράμματα βρίσκονται από πίσω. Σκέφτηκα να πούμε education for all, εκπαίδευση για όλους, γιατί αυτό δείχνει περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι εκπαίδευση για όλους οι δυνατόν με τα επιμέρους υποπρογράμματα. Τέλος πάντων θα έχουμε καιρό για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Α, να προσθέσω μία παρατήρηση ακόμη. Στις τις δραστηριότητες Ζαν Μονέ. Ε, εδώ μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να κινούμεθα στην αγορά. Ε, αυτοί, αυτά τα προγράμματα και αυτοί οι φορείς πάντοτε είχαν μεικτή χρηματοδότηση. Δηλαδή ε, λειτουργούσαν στην αγορά επιχορηγούμενοι. Ε, δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε την ύπαρξή τους όμως. Ε, και γι' αυτό να μην ε, ε, ε, τονίσουμε ιδιαίτερα την συνιστόσα της αγοράς. Συμφωνώ δηλαδή από αυτού με την πρόταση της Ντόρης. Ευχαριστώ. Μάρκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Ελπίζω να μην προσληθεί η Κομισιόν που θα πω ότι αυτή η πρόταση μου φαίνεται πολύ πιο κατανοητή, πιο ορθολογική από εκείνη που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το έρασμος για όλους, μας λέγατε ότι υπήρχαν τρία προβλήματα βασικά. Το πρώτο ήταν το, λέγαμε μάλλον, ότι ήταν τρία τα προβλήματα. Καταρχάς το όνομα. Σήμερα ακούμε ότι το έρασμος είναι ένα γνωστό και σημαντικό όνομα, αλλά όπως είπε και η κυρία Τρούπελ, παραπλανητικό, γιατί περιορίζεται σε ένα τομέα το Εράσμους. Εδώ στο Εράσμος βλέπω τόσους καθηγητές, τόσους μαθητές, τόσους φοιτητές που έρχονται εδώ μέσω άλλων προγραμμάτων. Να κρατήσουμε λοιπόν όλες τις ονομασίες που υπάρχουν. Και το Εράσμος μην ξεχνάμε ότι υπάρχει, είναι γνωστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, το ψάξουμε. Ε, αλλά βεβαίως πρέπει να ξέρουμε ότι το, το Erasmus for All δεν είναι το καλύτερο δυνατό όνομα. Επίσης, εμείς ξεκινήσαμε από την ιδέα να μοιράσουμε τα δύο προγράμματα. Θέλαμε τη διάκριση ανάμεσα την εκπαίδευση από τη μία και την ε, νεότητα και τον αθλητισμό από την άλλη. Υπάρχει τώρα αυτή η ενδιάμεση πρόταση. Το βασικό ήταν να κρατήσουμε μια σαφή ταυτότητα της νεολαίας και του αθλητισμού μαζί με την εκπαίδευση και στην έκθεση αυτή αυτό προκύπτει ξεκάθαρα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι απέναντι σε αυτό το θέμα και η Κομισιόν. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι απαραίτητο να κρατήσουμε διαιρεμένες τις τρεις ενότητες με ένα προϋπολογισμό για τις εθνικές υπηρεσίες. Και εδώ θα πρέπει να δούμε τι λειτουργεί και να το κρατήσουμε. Σίγουρα σε ορισμένες ε, χώρες Μία είναι η υπηρεσία. Εμείς ε, στην Ιταλία έχουμε δύο, γιατί αυτό βοηθάει και τη διάδοση, αλλά και την προσφορά υπηρεσιών για τα θέματα που μας απασχολούν. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να αναγκάσουμε τους πάντες να έχουν μία υπηρεσία. Φυσικά ο προπολογισμό θα είναι δεδομένος και θα πρέπει να το σεβαστούμε τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία ήταν τα πιο επικριτικά στην ε, έκθεση της ε, Doris Pack ε, νομίζω ότι προτάσσονται πολύ καλά, εξηγούνται πολύ καλά. Κάποια άλλα θέματα, αρκετά σημαντικά, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για τα, τους φορείς, τα Ινστιτούτα Ζαμονέ. Αυτή η διάκριση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και να είναι υπερητή. Ε, στο εσωτερικό των κρατών μελών. Και το τελευταίο είναι των πόρων. Θα ήθελα, μια και είμαστε εδώ το Κοινοβούλιο, που θα θέλαμε να αποφασίζουμε κι εμείς για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα κονδύλια. Μαζί με τους πολύ ικανούς και χρήσιμους υπαλλήλους, αλλά το κοινοβούλιο πάνω απ' όλα θα πρέπει να αποφασίζει πώς διαχειριζόμαστε τα διαθέσιμα κονδύλια. Και νομίζω ότι και αυτό το θέτει ε, το, το, προτάσει η, η έκθεση Doris Pack. Δίνει έμφαση σε αυτό. Ευχαριστώ κυρία Κάμαρβερτ. Ευχαριστώ Ντόρις και για την παρουσίαση της έκθεσης. Προσυπογράφω όλα όσα είπες και δεν θα τα επαναλάβω. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και με ενοχλεί στην πρόταση της Κομισιόν είναι ακριβώς αυτό το θέμα ότι όλα τα ανάγουν στην οικονομική χρησιμότητα παραλείποντας την κοινωνική ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη. Νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουν αυτό. Όσο ωραία και πολύτιμα να είναι, και αν είναι τα προγράμματα, δεν είναι προγράμματα που θα, που θα καταπολεμήσουν την οικονομική κρίση. Άλλωστε δεν έχουν πρικοδότηση τέτοια που θα τους επιτρέψει αυτό, ούτε μπορούν να καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Αυτά είναι πρόσθετα προγράμματα που δίνουν στους νέους και, τους, και στους ε, μεγαλύτερους ανθρώπους την δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό, να μάθουν εκεί, να αποκομίσουν εμπειρίες από εκεί, μια συμβολή στην ανέλξη της προσωπικότητας, ε, να συμβάλλουν ε, σε όλα αυτά. Δεν μπορεί όμως να καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων και την οικονομική κρίση. Το λέω αυτό για να μην έχουμε λάθος προσδοκίες από το πρόγραμμα που δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και ούτε πρέπει άλλωστε αφού η στόχη του είναι διαφορετικοί. Γι' αυτό με ενοχλεί επίσης ότι εν μέρη η συζήτηση για το όνομα έχει κάνει μια ζημιά. Ε, είχα τελευταία καλέσει μια σχολική τάξη και τη δασκάλα τους που είπε ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε στο μέλλον να, κάνουμε, να συμμετέχουμε σε προγράμματα στο Κομένιους. Και είπε, ε, βιαστείτε όμως γιατί το πρόγραμμα δεν θα υπάρχει σε δύο χρόνια. Ακριβώς αυτές οι συζητήσεις κάνουν κακό. Και ήδη από τώρα γίνεται ζημιά μετά τις προτάσεις της Κομισιόν και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τέτοιε υποθέσεις δεν πρέπει να εδρεωθούν στον πληθυσμό ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό η πρόταση που έκανε ε, είναι πολύ καλή. Να γίνει σαφής υποδιέρεση, ε, νεολαία, αθλητισμός, εκπαίδευση, να έχουμε το σαφή διάρθρωση των προγραμμάτων, να διατηρήσουμε τα παλιά ονόματα και έτσι να είναι σαφής η στόχη. ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Δηλαδή, ποια προγράμματα μπορούν να αξιοποιήσουν, από πού μπορούν να ωφεληθούν, γιατί τώρα όλα αυτά είναι συγκεχημένα και στο τέλος δεν νιώθει κανείς ότι έχει κάποιο κομμάτι του προγράμματος νόημα για εκείνον ή για εκείνην. Πρέπει λοιπόν εδώ στην Επιτροπή να μιλήσουμε με μια ενιαία φωνή και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, ελπίζω ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλά προοικοδοτημένο πρόγραμμα που θα έχει σαφείς δομές, σαφείς γραμμές στον προϋπολογισμό για να ξέρουμε τι ε, διατίθεται και τι δεν διατίθεται. Περιμένω με χαρά την επόμενη συζήτηση στο μέλλον. Η Μαρή Τερέζ. Ευχαριστώ για αυτή την πλήρη και ακριβή ανάλυση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έρασμος για όλους. Συμφωνώ και προσυπογράφω τη συζήτηση για τον τίτλο. Η εκμάθηση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου είναι κάτι πολύ πιο γενικό και θέλει να καλύψει όλα τα στοιχεία, όλες τις πλευρές που καλύπτει αυτή η πολιτική το όνομα έρασμος είναι πολύ γνωστό, αλλά περιοριστικό. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά και αναφέρθηκαν. Η αντάλλαγη καλών πρακτικών, η δικτύωση μεταξύ σχολείων, ε, πολυμερή προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα στα κράτη-μέλη. Τα υπάρχοντα προγράμματα ε, είναι γνωστά και αναγνωρίζονται, έχουν αρκετή ορατότητα. Το είπαν όλοι οι ομιλητές. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την ορατότητα ούτω ώστε να γίνονται κατανοητοί οι στόχοι μας. Επίσης, αυτές οι προτάσεις της ε, Κομισιόν έχουν μια κάποια στρατηγική, βασίζονται σε μια κάποια αξιολόγηση και αν ναι, ποια είναι, θα θέλαμε να τη μάθουμε. Αναλύονται οι ανάγκες, γίνονται κάποιες διαπιστώσεις. Ε, αυτά τα προγράμματα λειτουργούν καλά, γιατί να τα αλλάξετε, να τα καταργήσετε προσπαθούμε να βρούμε τη λογική και θέλουμε να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνεκτικότητα. Την ψάχνουμε λοιπόν. Συμφωνώ και με το συμπέρασμα της Ντόρης ότι είμαστε πολιτικοί. Εμείς αποφασίζουμε για τις στρατηγικές. Εμείς αποφασίζουμε για τον προϋπολογισμό γιατί έχουμε την αρμοδιότητα γι' αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε και αυτή η πρόταση της Κομισιόν δεν θα πρέπει να έρχεται ενώπιόν μας μόνο και μόνο για να την επικυρώσουμε. Έχουμε να κάνουμε προτάσεις και χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει ομοφωνία εδώ μεταξύ μας. Υποστηρίζουμε λοιπόν όλα όσα μας παρουσίασες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σχηματικό εδώ, να είμαι σύντομο, γιατί νομίζω ότι υπόθηκαν όλα. Καταρχήν θέλω να επιμείνω επί του ονόματο. Πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλο λάθο να δώσουμε αυτό το όνομα στο πρόγραμμα για δύο λόγους. Ε, καταρχήν ε, γιατί δεν είναι κατάλληλο για το ίδιο το πρόγραμμα, δεν λέει τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και επειδή δημιουργεί σύγχυση για το πρόγραμμα Εράσμους ε, και για αυτούς τους δύο λόγους νομίζω ότι θα έπρεπε να διατηρηθούν ε, οι υπόλοιπε ονομασίες που ανέφερες ε, γιατί είναι κάτι που γνωρίζουμε ήδη και κοστίζει πάρα πολύ στον εμπορικό κόσμο να καταργούμε μια επισήμανση και θα ήταν κρίμα εδώ να χάσουμε αυτούς τους τίτλους σε ό,τι φορά τώρα τον αθλητισμό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ε, μικρό κομμάτι του αθλητισμού ε, εδώ, όμως ε, παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ουσιαστική αύξηση των πόρων για τον αθλητισμό και δεν προσφέρεται ε, κάποια οικονομική υποστήριξη σε θέματα οριζόντια όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα για τον Αθλητισμό, η Ευρωπαϊκή Μέρα για τον Αθλητισμό, η προώθηση των αυτόχθονων ε, σπορ, δηλαδή που ε, ουσιαστικά τα βρίσκουμε σε διάφορες χώρες και αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ό,τι αφορά τις δραστηριότητες Ζαν Μονέ. Εγώ δεν ε, είμαι υπέρ ε, των ονομαστικών επιχορηγήσεων. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να υποστηρίξουμε τα εφιστάμενα προγράμματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται και επικαιροποίηση. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι τα προγράμματα θα πρέπει να γίνονται μέσω ονομαστικών δεν θα πρέπει να είναι ονομαστικά προγράμματα που θα αναθέτονται έτσι. Και για το θέμα του προπολογισμού ε, αναφέρθηκε μια αύξηση 70% είναι λίγο αλλά και πολύ ταυτόχρονα έτσι λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω σε ποια κεφάλαια σκέφτεστε ε, να υπάρχει αυτό το 70% και εμείς ε, ως Κοινοβούλιο να είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε πού θα γίνει αυτή η αύξηση και πού θα πάει αυτή η ποσότητα, αυτό το ποσό κατά τα λοιπά. Συμφωνώ με τις προτάσεις σου. Ευχαριστώ. Κέκοπ. Thank you very much, uh, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ γνωστό το πρόγραμμα Erasmus ε, και ε, λέγαμε όταν ε, ε, έχω χρήματα το 1950 λέγαμε όταν θα έχω χρήματα θα αγοράσω βιβλία και αν μου μείνουν θα αγοράσω ρούχα εδώ ουσιαστικά πρέπει να δούμε τους όρους αναφοράς ε, του Εράσμους και ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα θέματα που θα θέσουμε σε προτεραιότητα. Εγώ μιλώ ε, και εκ μέρους του αυτού μου εκπροσωπώ και την κυρία Άννα Μακλάρκ και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το μέγεθος του προπολογισμού και πιστεύω συγκεκριμένα όχι μόνο για το μέγεθος του προπολογισμού αλλά και για το ότι το 40% αυτού δεν ε, έχει εγγραφεί σε συγκεκριμένη προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν, ε, αν ε, κάνουμε γενικά πράγματα με τον προπολογισμό, τότε γενικά δημιουργούμε πολλά προβλήματα και δεν έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Έχουμε ανησυχίες για το σύστημα του Μάστερ και θέλουμε να υπάρχει προσθεμένη αξία και θέλουμε να δούμε και πώς θα λειτουργήσει ε, υπάρχουν ε, και τα θέματα του ελέγχου και μπορεί να προκύψουν κάποιε δυσκολίε. Ε, και εγώ το ξέρω γιατί έχω υπουργική εμπειρία στο Ρωμένο Βασίλειο με διάφορε τέτοιε επιχειρήσει για τα προγράμματα Ζαν Μονέ που λαμβάνουν 78 εκατομμύρια ευρώ Νομίζω ότι η κύρια χρηματοδότηση είναι κάτι και το οποίο θα πρέπει να στρεφόμαστε κατά. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρατηρήση σας κυρία Πρόεδρε και συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω ότι ε, πάντοτε θεωρούσαμε ότι αν το Εράσμος θα πρέπει να κάνει κάτι θα ήταν να ενθαρρύνει τους νέους. Όπως ε, είπατε, έχουμε και το θέμα της απασχόλησης. Θα έπρεπε τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα ε, επικεντρώνεται στην υποστήριξη της βάσης και ας απευθυνθούμε στους νέους Ευρωπαίους πολίτες ε, που βρίσκονται σε ανάγκη και νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ καλό. Το πρόγραμμα του αθλητισμού είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλή ευκαιρία. Πρέπει να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι νέοι καθώς ε, είναι το μέλλον της Ευρώπης ε, και δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε στους ε, μεγαλύτερους ηλικία και επίσης για το μη εμπορικό, η μη εμπορική διαφημίση νομίζω ότι θα πρέπει να συνεισφέρει και η βάση θα πρέπει ε, να συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί, να γνωριστούν οι νέοι μεταξύ τους ε, και να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των νέων στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αντί να έχουμε μπλοκ ε, πέντε οργανώσεων σε τρεις διαφορετικές χώρες, θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε την εμπλοκή περισσότερων τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων, τον ίδιο τρόπο με τα προγράμματα leaders στην ανάπτυξη της υπαίθρου που νομίζω ότι είναι ε, πολύ ικανοποιητικά. Το να εμπλέξουμε ε, τη βάση, το να συμμετέχουν οι νέοι, να επικεντρωθούμε σε αυτά που αφορούν τους νέους ε, είναι κάτι που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρτιν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που έγιναν ε, στην εισαγωγή σας και πιστεύω ότι πολλοί τοποθετήθηκαν επί του θέματος αυτού. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να παρουσιάσουν περισσότερες δυσκολίες για το να καταλήξουμε σε συμφωνία σε αυτήν την Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Συνολικά πιστεύω ότι είναι καλή η πρόταση της Κομισιόν, συμπεριλαμβάνει πολλά στοιχεία από το προηγούμενο πρόγραμμα κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την απλούστευση και το streamlining ε, και αυτά υποστηρίζουν και υπόλοιπε ομάδες. Όμως θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερις ε, τομείς της πρότασης που νομίζω ότι μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά το Κοινοβούλιο. Καταρχήν, το πιο ενδιαφέρον θέμα φαίνεται να είναι η ονομασία η επλούστευση προκάλεσε μεγάλη σύγχυση σε πάρα πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ακούσαμε ήδη. Και πράγματι δεν είναι απολύτως σαφές που εμφανίζονται το θέμα της επαγγελματικής ε, κατάρτισης ε, στην πρόταση. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Επικοδομητικά συμφωνώ με την Κομισιόν ότι το, είναι, ε, το όνομα Εράσμος είναι πολύ ισχυρό και πολύ γνωστό και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με φιλόδοξο τρόπο. Λεχθέντος αυτού είναι σαφές ε, ότι ε, και ε, τα ονόματα Κομίνιος και Λεωνάρντο είναι ισχυρά. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε σε έναν κατάλληλο συμβιβασμό για το θέμα αυτό και ενυπομονώ να δω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία για το θέμα της νεολαίας, για το κεφάλαιο της νεολαίας. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε πολλά κεφάλαια. Η νεολαία πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Και για τον αθλητισμό, το στοιχείο του αθλητισμού αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν και φυσικά είναι κάτι σκόπιμο και σχετικό. Θέλω να τονίσω τη σημασία της προώθησης της υγείας μέσω της σωματικής δραστηριότητας. Τα κράτη-μέλη θα εξοικονομούσαν πολλά χρήματα αν ε, γυμνάζονταν περισσότερο οι πολίτε και τώρα λαμβάνουν χώρα πολλέ δραστηριότητε. Νομίζω ότι πρέπει να τι υποστηρίξουμε και να βρούμε και τι κατάλληλε ιδέε περί δραστηριοτήτων. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε ιδέε ήδη, πρέπει να τι υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά τι δράσει Ζαν Μονέ ε, και την υποστήριξη για τα ιδρύματα, θα συμφωνούσα ότι είναι παράξενη αυτή η απόφαση να προωθήσουμε δύο και όχι τα έξι εξ αυτών. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ε, γιατί έχει ληφθεί αυτή η θέση, όμως εγώ θα πρότεινα να υποστηρίξουμε και τα έξι. Γιατί δεν είναι λογικό κατά την άποψή μου πλέον να υποστηρίξουμε τα δύο ιδρύματα και όχι το σύνολο των ιδρυμάτων. Έτσι λοιπόν αυτό θα ήταν το σημείο εφετηρίας μου τη συζήτηση αυτή. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Μπάγκο. Μην επαναλάβετε αυτά που είπαν οι άλλοι. Καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν που περιλαμβάνει και τον αθλητισμό στις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές οι δράσεις ε, για τον αθλητισμό συνάδουν με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Οι προτάσεις είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς, όμως το τμήμα της εφαρμογής ε, περιγράφεται με πολύ γενικούς όρους και δεν ε, βλέπω πώς θα εγγυθεί η συνέχιση των προγραμμάτων στη συνέχεια σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για την νεολαία. Νομίζω πρέπει να αλλάξει και το περιεχόμενο, όχι μόνο η μορφή. Σε ό,τι αφορά την διαβίωμαθησή Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τμήμα του προγράμματος, αλλά δεν είναι ο μόνος στόχος του προγράμματος αυτός η διαπολιτισμική μάθηση δεν θα αποτελούσε τμήμα του σημερινού προγράμματος έτσι όσο έχει αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν θα υποστήριζα και η νεολαία να μπει σε καθένα κεφάλαιο του προγράμματος και για τις δράσεις Ζαν ε, Μονέ. Το Συμβούλιο έλαβε μια σχετική απόφαση, όμως αυτό δεν με δεσμεύει ως ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι λοιπόν υπέρ των όσων είπατε και εσείς Πρόεδρε ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να δοθούν βάσει αιτήσεων. Κάτι τέτοιο θα προωθούσε και τον ανταγωνισμό και θα βελτίωνε την ποιότητα των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν δεν βλέπω κανένα λόγο να ε, αναφέρουμε σε κατάλογο αυτούς, τους, ε, αυτά τα ιδρύματα. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε αυτό κι άλλο. Η Ζαμπίνε, πολύ σύντομη θα είμαι, συμφωνώ με πολλά και με τη βασική προσέγγιση του εγγράφου όπως παρουσιάστηκε. Νομίζω ότι συνιστά τη σωστή κατεύθυνση και η διατήρηση του παλιού ονόματος ε, αυτά που είπαμε με βρίσκει σύμφωνη. Όταν ρωτήσω τα, τους μαθητές του Κομένιους, ε, όσοι γνωρίζουν το Κομένιους δεν ταυτίζονται με το Εράσμους. Είναι διαφορετικό. Ε, βλέπω ότι υπάρχουν περισσότεροι εκπρόσωποι της Κομισιόν ε, σήμερα το απόγευμα από ό,τι το πρωί. Και ε, θα ήθελα να ρωτήσω, όταν προτείνει 56% η Κομισιόν, και το 44% να είναι ευέλικτο χρήμα, ας πούμε, με αυτό το διαχωρισμό τι έχει υπόψη της. Κάποιο σκεπτικό θα πρέπει να έχει. Τα 44% δηλαδή τι σκοπεύει να τα κάνει η Κομισιόν. Γιατί όταν τα χωρίζει έτσι, κάπου πρέπει να το στηρίζει αυτό. Πολύ θα με ενδιαφέρει μια απάντηση από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, εσείς, ε, από την Κομισιόν, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, γραφειοκράτης, και ελπίζω να είμαι από τους ε, πολύ καλούς, από τους υπέροχους, δεν θα μιλήσω για συναισθήματα, αλλά για το τι θα πρότεινα και εδώ έχω την αισθησία ότι στα περισσότερα σημαντικά θέματα συμφωνούμε. Συμφωνούμε για τη σημασία τη παιδεία, τη εκπαίδευση και τη νεολαία. Συμφωνούμε γιατί είναι σημαντικό να συνδέσουμε καλύτερα το πρόγραμμα με τι ε, προτεραιότητε πολιτική. Επίση συμφωνούμε για την ολιστική προσέγγιση, δηλαδή την προσέγγιση που θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ε, άτυπη και την επίσημη εκπαίδευση και επίσης συμφωνούμε επί της απλούστευσης. Και τέλο πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε για τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν κάποια σημεία όπου νομίζω ότι ακόμα και αν φαίνεται ότι διαφωνούμε, μάλλον πρόκειται περί παρεξήγησης. Δηλαδή δεν ήμασταν αρκετά σαφείς στην πρότασή μας. Αυτό σημαίνει. Θα αναφέρω τρία-τέσσερα σημεία. Καταρχήν, η σημασία που προσδίδουμε στην νεολαία. Φυσικά προσδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην νεολαία. Συμφωνούμε με όλους όσους λένε, μεταξύ μόνο συγκεκριμένα, ότι η απασχόληση και η είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και ακριβώς ε, γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η ολιστική προσέγγιση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε μαζί μας το ότι αν αντιμετωπίσουμε ε, την πρόορια εγκατάλειψη του σχολείου είναι σημαντικό για τις ευκαιρίες που θα έχουν οι νέοι. Και επομένω να αντιμετωπίσουμε όλε τι πτυχέ που σχετίζονται με την νεολαία, είτε στην επίσημη είτε στην ε, άτυπη εκπαίδευση, είναι κάτι σημαντικό. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να αφήσω εδώ έχει να κάνει με κάτι που θεωρήσατε ως ε, οικονομική προσέγγιση της πρότασης αυτής, ορισμένη από εσάς. Ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν λέμε ότι συνδέουμε το πρόγραμμα αυτό με το εφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής, δηλαδή με το πρόγραμμα για την εκπαίδευση και κατάρτιση για το 2020, που περιλαμβάνει και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, όπου έχουμε και εκεί σημαντική κοινωνική διάσταση και μια σημαντική πτυχή ενεργού συμμετοχή των νέων και πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Και ακριβώ για αυτό το λόγο, για πρώτη φορά βάλαμε αυτέ τι αναφορέ ε, στην πολιτική ω κύριου στόχου του προγράμματο ε, και προ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα καλύπτει όλου του πολύπλοκου ε, τομεί των δράσεων στον τομέα τη εκπαίδευση, τη νολέα, του αθλητισμού κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε περαιτέρω δουλειά να κάνουμε για να εξηγήσουμε καλύτερα τι κάνουμε. Και ένα άλλο θέμα παρεξήγηση ε, είναι το επίπεδο τη λεπτομερού περιγραφή των δράσεων. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την πρότασή μα, βλέπουμε το ίδιο επίπεδο λεπτομέρεια, εκτό από το ότι δεν περιγράφεται με τον ίδιο τρόπο στου διάφορου τομεί. Δηλαδή, αν δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Στον τομέα της κινητικότητας στην εκπαίδευση, και θα αναφέρω την πρότασή μας, λέμε ότι θα έπρεπε να υποστηρίξουμε την διασυνορική κινητικότητα των ε, φοιτητών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών ε, και η κινητικότητα αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή ε, σπουδών σε ένα άλλο ίδρυμα κτλ. Και ακριβώ αυτό λέμε εδώ και πιθανόν αυτό θα λέμε και στο σημερινό πλαίσιο έτσι λοιπόν, αν δείτε τι προτείνουμε, θα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει περισσότερη σύγκληση. Όμως, όπως είπατε και εσείς, κυρία Πάρκα, εδώ μιλάμε μεταξύ πυρογνωμόνων. Και αυτό είναι καλό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είναι καλέ και αποφάσει. Όμω τι σημαίνει ότι ξέρουμε πολλά ε, για όσα κάνουμε σήμερα από το σημερινό πλαισίο και πολλά από τα πράγματα που κάνουμε είναι καλά και γι' αυτό προτείνουμε να τα προωθήσουμε. Αλλά πολλέ από αυτέ τι λεπτομέρειε δεν υπάρχουν στη νομική βάση υπάρχουν ε, στα σχετικά εγγραφά εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, ε, θα ήταν να συγκρίνουμε όμοια πράγματα, να συγκρίνουμε τη σημερινή νομική βάση, όχι τι καθευτηρίε γραμμέ για την εφαρμογή, όχι την εφαρμοστική απόφαση, αλλά τη βάση LB με την βάση για το Erasmus για όλου. Και βέβαια δεν μπορεί να έχουμε μόνο καλά νέα, νομίζω ότι υπάρχουν και ορισμένα σημεία όπου αποκλίνουμε κάπως το πρώτο επί του τίτλου, επί της ονομασίας. Και άκουσα πολλούς να λένε ότι αυτή η ονομασία δεν είναι κατάλληλη και κάποιοι είπαν ότι αυτό το όνομα είναι το κατάλληλο. Φυσικά θα στραφούμε σε εσάς και πάλι και στο Συμβούλιο για να λάβουμε την τελική απόφαση. Όμως υπήρξε μια σαφής ανάλυση της κατάστασης, όχι μόνο σε αυτό, το θέμα, αλλά και σε όλες τις προτάσεις ε, και σίγουρα είδατε την μελέτη αντικτύπου και θα είδατε πώς εξηγούμε τις επιλογές μας. Για το Εράσμους, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, ε, το καλύτερο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, και νομίζω ότι είναι καλό να κατομίσουμε πάνω σε αυτό το σήμα για να δυσφαλίσουμε ότι προβάλλεται το πρόγραμμα αυτό επαρκώς, καθώς αποτελεί επιτυχία. Και ε, ακόμη και αν ε, το Κοινοβούλιο παρουσιάσει νέα πιλωτικά προγράμματα, αν κάνω λάθος, ε, υπήρξε ένα πρόγραμμα που παρουσίαση το Κοινοβούλιο που λέγεται Εράσμους για τους μαθητευόμενους. Και φυσικά αυτό το εμπορικό σήμα, αυτή η ονομασία μπορεί να βοηθήσει να γίνει πιο γνωστό το πρόγραμμα. Το άλλο θέμα, στο οποίο διαφωνούμε, είναι η ευελιξία. Αυτό που προτείνουμε δεν είναι ακριβώ 56%, πρέπει να προσθέσουμε και το 5% για τη διοίκηση. Έτσι λοιπόν φτάνουμε περίπου στο 60%. Προτείνουμε ε, να ενεργοποιηθεί από τον προπολογισμό και προσπαθούμε σήμερα να εκτελεστεί από τον προπολογισμό προσπαθούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε για τις προτεραιότητες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 2019 και το 2020. Έτσι λοιπόν, ε, καλό θα είναι να συζητήσουμε τον καθαρισμό των προτεραιοτήτων ε, και να έχουμε ελάχιστη εκταμείευση ένα τομέα και να καταστήσουμε δυνατό αφετέρου ότι θα έχουμε οριζόντιες προτεραιότητες που θα καλύπτουν το τομέα των σχολείων και της νεολαίας, το τομέα της νεολαίας ή της ε, διαβίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης ή άλλες οριζόντιες δραστηριότητες. Και κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, για την ε, διαχείριση. Νομίζω ότι η διαχείριση ενός τέτοιου προγράμματος είναι πολύ σημαντική και καθώς θα έχουμε ομοιόμορφους κανόνες, θα είναι σημαντικό οι δράσεις που προτείνουμε να είτε είναι η κινητικότητα, η στρατηγική συνεργασία, είτε η υποστήριξη τη πολιτική να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε κράτο μέλο. Ή τουλάχιστον να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο μέσα σε ένα κράτο μέλο, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να ε, διευκολύνουμε τη ζωή όσων ωφελούνται των δικαιούχων, ε, είναι σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα διαχείριση ε, το οποίο θα εφαρμόζεται συνεπώ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Κορέλ. Πρόεδρος είμαι, πρέπει να είμαι προσεκτική. Αγαπητέ κυρία Κορέλ, διαπιστώσατε, διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένα πράγματα συμφωνούμε, καλά λέτε, σε άλλα δεν συμφωνούμε με χαρά διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν τους πειράζει ο τίτλος. Δεν λέω, αλλά οι περισσότεροι δεν συμφωνούν. Δεν πρόκειται για τον τίτλο. Δεν επιμένω να αποδείξω ότι εγώ έχω δίκιο. Όλοι το εξήγησαν και εγώ το εξήγησα. Είναι παράλογο, είναι παραπλανητικό, δημιουργεί σύγχυση, δεν λέει αυτό που θέλουμε. Προσοχή λοιπόν. το Κοινοβούλιο είχε πει ότι θέλουμε εράσμου και για του μαθητευόμενους, αλλά δεν μπορεί να βασιστούμε εκεί. Και μάλιστα τους είχα πει, το Λεωνάρδο δεν το ξέρετε, αυτό είναι το εράσμους για τους μαθητευόμενους. Αν δεν το ξέρετε ω βουλευτέ, πώς κάνετε αυτή την παράδοξη πρόταση που τώρα την παίρνει η Κομισιόν σαν μπούμερα. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, δεν θέλουμε πάλι να ξαναπιάσουμε το θέμα. Συμφωνούμε στην απλοποίηση, απλούστευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απλουστευτεί και η διαδικασία υποβολής προτάσεων. Όχι μόνο εδώ και στο Creative Europe παντού υπάρχει πρόβλημα. Ούτε είναι μόνο πρόβλημα της Κομισιόν αυτό. Είναι πρόβλημα διοργανικής συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που θέλουν να τα ελέγχουν όλα μέχρι τελευταίου κόμματος. Τα χρήματα που δίδονται εδώ στο Κομμένιο, στο Λεωνάρντο δεν είναι ε, λεφτά για να πλουτίσει κανείς, όμως χρειάζονται από τους ετούντες. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε προς το συμφέρον των συμμετεχόντων να πλουστεύσουμε το πρόγραμμα. Γι' αυτό είναι παράδοξο που παρά τις δύσκολες ε, διαδικασίες υποβολής εκπλήσει ότι απορροφήθηκαν όλα τα χρήματα αυτού του προγράμματος. Άλλο παράδειγμα τέτοιο δεν υπάρχει από το, το κοινωνικό ταμείο, τα διαφορετικά ταμεία, δεν απορροφώνται 100% τα κονδύλια, ενώ εδώ ναι. Και είναι σαφές και νομίζω και η κυρία Τρούπελ το είπε προηγουμένως, ότι τα θεσμικά όργανα, όχι, τα ιδρύματα που προωθούμε Πρέπει να βρουν και άλλα κονδύλια για να επιβιώσουν. Το, η Μπρούζ, το Μάστριχτ δεν μπορούν να βασιστούν και να ζήσουν μόνο με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι σημαντικά. Το, το, η η Τρίερ, το Μάστριχτ είναι παιδιά αυτού του κοινοβουλίου. Ιδέες δηλαδή που πήραν σάρκα και οστά. Και οι συνάδελφοι που λένε «Ε, δεν πρέπει να συνεχίσουμε να τα στηρίζομαι. Σε αυτούς απαντώ ότι δεν πρέπει να επανεφευρίσκουμε τον τροχό συνεχώς. Κάτι που έτρεξε τόσο καλά επί δεκαετίες, δεν μπορώ τώρα εγώ ξαφνικά να το καταργώ. Παρακαλώ θερμά λοιπόν σε αυτό το τομέα ε, να συμφωνήσετε μαζί μου ή όλοι ή τίποτε. Και αν δεν είναι κανείς, όπως λέει ο κύριος Μπάγκο, τότε όλοι θα πρέπει να ε, υποβάλουν προγράμματα για να πάρουν χρήματα. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο δαπανήρη διαδικασία. Μεγαλύτερη διαχείριση, πιο πολλέ διοικητικέ δαπάνε από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που εδώ και μερικές βδομάδες ε, εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα. Κάναμε και εντατική ανταλλαγή απόψεων. Ε, δεν θέλω να επιβάλλω την απόψή μου και να δικαιωθώ. Εγώ ήμουν ευγνώμων για το πρόγραμμα Lifelong Learning όταν ήρθε και ήθελα να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τη διαδικασία, όχι το όνομα εδώ. Και συμφωνώ με την Κομισιόν και έτσι θα προχωρήσουμε. Για τον αθλητισμό, κυρία Κύρκοπ, να το συζητήσουμε αυτό, αλλά οπωσδήποτε αυτό το θέμα θα τεθεί όταν περάσουμε στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλά, πολλές προτάσεις για το Εράσμους και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πλαίσια. Πάντως πέρασε το μήνυμα. Για τους εθνικούς οργανισμούς, οι εθνικοί οργανισμοί λειτουργούν, αλλά αυτό που χρειάζονται είναι ε, ένα πόρταλ κοινοτικό να παρουσιάζει όλα τα προγράμματα όταν πάμε στο Κομένιους για παράδειγμα. Τώρα η Κομισιόν ασχολείται για να κάνει κάτι τέτοιο για το παλιό πρόγραμμα και θα έχουμε και το καινούριο πρόγραμμα, ελπίζω, με το παλιό του πρόγραμμα. Αν έχει κανείς μια πρόταση άλλη, καλύτερη από το lifelong learning, κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να είναι εξίσου καλή πρόταση όπως το lifelong learning. Α, ξέχασα, Έχουμε εκπροσώπηση του Συμβουλίου. Κυρία Άντερσεν, σας δίδω το λόγο για να μας πείτε γρήγορα τι πιστεύει το Συμβούλιο, τι ενέκρινε, τι απέρριψε. Κυρία Άντερσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τη δουλειά που κάνει το Συμβούλιο επί του προτινόμενου προγράμματος κατά τη διάρκεια της Ανικής Προεδρίας. Φυσικά σεβόμαστε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία και ακριβώς γι' αυτό περιμένουμε την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ως Προεδρία έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση ε, στη διαπραγματεύση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τις ε, νομικές πράξεις και ε, το πρόγραμμα αυτό Θέλουμε να το συμφωνήσουμε. Αυτό συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα που προτείνεται. Αυτή τη μερική γενική συμφωνία την πετύχαμε στις 11 Μαΐου στο Συμβούλιο Υπουργών. Είναι μερική η συμφωνία γιατί περιμένουμε την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Είναι μερική όμως γιατί δεν περιλαμβάνει τις σχέσεις, τα στοιχεία που αφορούν τον προϋπολογισμό και, ή τους άλλους κανονισμούς που τους διαπραγματευόμαστε σε άλλα μορφώματα, παραδείγματο χάρη τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η μερική γενική ε, συμφωνία ε, είναι υπέρ της απλουστευμένης, ολοκληρωμένης ε, και ευρεία προσέγγιση κομισιών, εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός όλα μαζί. Κρατήσαμε την ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη του ενιαίου προγράμματος και της επίσημης και μη επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης, κρατώντας όμως και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα, όπως απεικονίζεται στο... και στα τρέχοντα προγράμματα. Οι διάφοροι τομείς και τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών έχουν τονιστεί στο κείμενο της ε, Μερικής ε, Γενικής Συμφωνίας, ε, παραδείγματος χάρη εκπαίδευση των υλίκων, ε, και ελάχιστες, ε, τα ελάχιστα κονδύλια για τους διάφορους τομείς που προτείνονται. Καθώς ε, αθλητισμός για όλους που έχει επίσης υπογραμμιστεί. Η διαβίου μάθηση είναι πιο προφανής αλλά από ό,τι στην αρχική πρόταση. Σε ό,τι αφορά αυτό το τμήμα της διαβίου κατάρτισης μάθησης πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την υποστήριξη για ένα ολοκληρωμένο ενιαίο πρόγραμμα και τις νέες δυνατότητες για να συνδέσουμε την επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση με τομή, ε, υπήρχε μια σαφής, ε, ένα σαφές αίτημα στο Συμβούλιο να προτάξουν περισσότερο το τομέα της νεότητας. Η συμφωνία ε, συμπεριλαμβάνει μια πρόταση για ένα ανεξάρτητο κεφάλαιο για την νεολαία και τη συμπερίληψη των ανοργάντων νέων ως ομάδα στόχος. Υπάρχουν τρία κεφάλαια δηλαδή, με τρεις γραμμές στον προπολογισμό. Ε, ο συμβασμός είναι ότι σε αυτή την γενική προσέγγιση ε, ο τομέας της νεολαίας έχει την ίδια, την ίδια διάρθρωση με τους άλλους τομείς, αθλητισμός κτλ. Ούτως ώστε να κρατήσουμε αυτά ωφέλη που θα είχαμε από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Άλλες αλλαγές που θα μπορούσαν να σε ενδιαφέρουν είναι ότι οι δείχτες έχουν φύγει από την νομική πράξη και θα αποφασίζονται στη στο πρόγραμμα της Επιτροπής, η οποία θα μπορεί να συνέρχεται σε διάφορες συνθέσεις. Τα κράτη-μέλη με βάση αυτή την ε, μερική προσέγγιση θα μπορούσαν να αποφασίσουν ε, τον τρόπο εφαρμογής που να είναι αποτελεσματικός ε, με σεβασμό της Ευρωπαϊκής Θεμοθεσίας και το Δημοσιονομικό Κανονισμό. Είναι σωστό ότι αυτή η μερική γενική προσέγγιση διέγραψε την αναφορά ή τις αναφορές σε ένα ενιαίο συντονιστικό φορέα η Εθνική Υπηρεσία στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πόσες υπηρεσίες ή φορείς θέλουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Και τα έξι ιδρύματα επίσης ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Ε, τελευταίο, η συμφωνία μας δεν προτίζει δεν προτείνει διαφορετικό όνομα από αυτό που προτείνει η Κομισιόν Έρασμος για όλους. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω ότι και τα τρία θεσμικά όργανα τελικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Ευχαριστώ και σε ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ είπα για τις τελευταίες μου λέξεις. Ευχαριστώ θερμά την Κομισιόν που θέλει να συνεργαστεί, το ίδιο και το Συμβούλιο, αλλιώς δεν θα υπήρχε πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η διαδικασία της συναπόφασης ε, και ε, όλοι προς την ίδια κατεύθυνση δρούμε και συνεργαζόμεθα δεν υπάρχουν διαφορές, λίγες είναι αυτές που έχουν μείνει και νομίζω ότι θα τις ε, διασκεδάσουμε και αυτές. Ευχαριστώ για την πρώτη συζήτηση. Θα έχουμε τον Ιούλιο δεύτερη συζήτηση και θα μπούμε πιο πολύ στις λεπτομέρειες των δομών. Είναι ε, πολλή δουλειά γιατί θα πρέπει με τις τροπολογίες μας, με τις προσθήκες μας να δούμε πώς θα τα ε, κάνουμε. Έχουμε και νομικό σύμβουλο. Χαίρομαι που θα έχουμε αυτή την καλή συνεργασία. Είναι δύσκολος ο φάκελος αυτός και πραγματικά χωρίς εσάς δεν θα τα καταφέρναμε. Ωραία. Θα λάβουμε υπόψη μας και αυτά που βρίσκουμε καλά στο θέμα, στο, στην πρόταση της Κομισιόν. Τελειώνουμε λοιπόν το ζήτημα αυτό και πάμε. Äh, Σημείο 12 θα πάμε, γιατί για τον προϋπολογισμό έχουμε τον συντάκτη της γνωμοδότησης εδώ και θέλει να θέσουμε το θέμα. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, Πρόεδρε για τη δική σας έκθεση «Έρασμος για όλους». Στις 19 Ιουλίου, στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές, θα ξανασυζητήσουμε το θέμα, όπου θα μπούμε πιο πολύ στις λεπτομέρειες του κάθε σημείου. Μετά τον Σεπτέμβριο στη συνεδρίαση θα υποβάλω εγώ την έκθεσή μου, το Σεπτέμβριο ε, κατά ένα μήνα το αναβάλαμε. Το Σεπτέμβριο θα υποβοληθεί η έκθεση. Θα έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες και τον Νοέμβριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Ε, έχει, έχει αναβληθεί, επειδή μεσολαβούν οι θερινές διακοπές. Εντάξει. Αντί να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο 11, θα πάμε στο 12, γιατί είναι εδώ ο εισηγητής από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Η Κομισιόν έχει σχέδιο προϋπολογισμού στις 24 Απριλίου, το υπέβαλε, για τον επόμενο χρόνο και υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που συνεχίζονται στον προϋπολογισμό. Πρώτο, ε, από τον προϋπολογισμό μας καλούν έναν αριθμό πιλωτικών προγραμμάτων και δράσεων να υποβάλουμε. Αυτό το κάναμε για να απαντήσει η Κομισιόν και πριν αποφασίσουμε να δούμε ποιες τροπολογίες θέλουμε να καταθέσουμε. Μετά έχουμε την γνωμοδότηση και ο συντάκτη της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Λόκεγκαρτ για να δούμε τι, προ... έχουμε στον προϋπολογισμό Και τέλος οι τροπολογίες ε, του προϋπολογισμού για το Συμβούλιο και το σχέδιο Προϋπολογισμού. Λοιπόν, Δίνω το λόγο στον κύριο Λάτφιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω κύριο Λαβία, που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να έρθω στην Επιτροπή Πολιτισμού για να σας μιλήσω για το, τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2013. Η διαδικασία για την έκριση του προϋπολογισμού είναι μακροσκελής. Ξεκίνησε με την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών το Μάρτιο στο Στρασβούργο από το Κοινοβούλιο. Παρουσιάσαμε ήδη και θα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια στενή συνεργασία με τις ειδικέ κοινοβουλευτικές επιτροπές, ούτως ώστε να εστιάσουμε στους πόρους και στις πρωτοβουλίες που αφορούν κυρίως ε, τις προτεραιότητες που έχει εντοπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ούτω ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή χορήγηση των ε, μικρών και, και ανεπαρκών πόρων. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες που διαλέξαμε για τον προϋπολογισμό του 2013. Ε, διανύουμε μια βαθιά κρίση και σε πολλά κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς θέλαμε τον προπολογισμό αυτό να τον, τον βασίσουμε στην ανάπτυξη από τη μία και στην απασχόληση από την άλλη και κυρίως στην απασχόληση των νέων πιο ειδικά. Αυτός ο προπολογισμό θα θέλαμε σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να εξεταστεί και να ερμηνευθεί με βάση αυτές τις προτεραιότητες. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι δύσκολο προπολογισμό, γιατί είναι ο τελευταίο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013. Ε, τα πρώτα χρόνια τη περίοδου προγραμματισμού είχαμε πολλέ ε, δεσμεύσει και τώρα σε αυτόν τον προπολογισμό έχουμε το πρόβλημα των πληρωμών. Τώρα εμφανίζεται. Επομένω, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με του πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα τι δεσμεύσει που είχαμε λάβει προηγούμενα χρόνια και αν τι καλύψουμε αυτέ τι δεσμεύσει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού ζήτησε αύξηση των δεσμεύσεων πληρωμών ε, επιπρόσθετων που φτάνουν στο 6,8% σε σχέση με τον προηγούμενο προπολογισμό. Σας είναι επίσης γνωστό ότι θέλουμε ότι για τους στόχους κατά προτεραιότητα εκεί να δώσουμε τους περισσότερους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτό θα το κάνουμε ε, σε όλες τις επιτροπές. Ένα σημαντικό στοιχείο που θέλω να τονίσω, βλέπετε και αυτή την έκθεση που μόλις μου μοιράστηκε και που αφορά τις, τα πιλωτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, αποφασίσαμε φέτος να υιοθετήσουμε μια διαδικασία που μας επιτρέπει να εντάξουμε στην τελική συμφωνία για τον προϋπολογισμό μόνο τις προτάσεις των πιλωτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων που είναι ε, εφαρμόσιμα. Γι' αυτό λοιπόν φτιάξαμε ένα χρονοδιάγραμμα που προβλέπει μέχρι το τέλος του μήνα την παρουσίαση στις επιμέρους επιτροπές, τις ειδικέ, τις, προτάσει προτάσεις για αυτά τα πιλωτικά έργα και προπασκευαστικές δράσεις. Αυτή η δουλειά εσείς την κάνετε, όπως βλέπω. Και αυτές οι προτάσεις θα περάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια πρώτη αξιολόγηση προκαταρτική για την σκοπιμόταν να προωθηθούν αυτές οι πιλωτικές δράσεις, ούτω ώστε μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουμε μια αξιολόγηση από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις δυνατότητες εφαρμογής αυτών των πιλωτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Αρχές ε, Σεπτεμβρίου, αν χρειαστούν, θα γίνουν οι προσαρμογές με τις απαραίτητες ε, προσαρμογές και αλλαγές. Και οι επιτροπές θα ψηφίσουν τις προτάσεις τους για πιλωτικά προγράμματα και προπασκευαστικές δράσεις. Με βάση τα περιθώρια που έχουμε στους επιμέλους τίτλους, στο τελικό πακέτο του προϋπολογισμού θα βάλουμε τις προτάσεις που θα προέρχονται από τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι θα βάλουμε μόνο εκείνες τις προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί ως εκτελεστές και εφαρμόσιμες. Γιατί σε μια εποχή λίγων πόρων, η να γελάδων, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δώσουμε πόρους για προγράμματα που δεν θα δουν ποτέ το φως. Γι' αυτό ακριβώς ε, υποβάλαμε αυτές τις προτάσεις πρώτα προς αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα εξετάσουμε μόνο και θα λάβουμε υπόψη μας μόνο αυτές που θεωρούνται εφαρμόσιμες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα προγράμματα που αφορούν τη δική σας Επιτροπή. Από την Επιτροπή περιμένουμε μία αξιολόγηση επί της ουσίας. Ζητάμε από κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αυτό το ζητάει πάντα Επιτροπή Προεπολογισμών. ε, ζητάμε να είσαστε ευαίσθητοι, ευαισθητοποιημένοι σε μια περίοδο κρίσης και δυσκολιών που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αξιολογήστε με προσοχή εκεί όπου θεωρείτε ότι μπορεί να είναι πιο χρήσιμη, χρήσιμο να δοθούν οι πόροι. Και ε, δέστε και ποιες είναι οι ενδεχόμενες αρνητικές προτεραιότητες, γιατί μπορεί να χρειαστεί να περικόψουμε. Καλό θα ήταν λοιπόν οι καθήλια αρμόδιε επιτροπέ να, έχουμε, να μας δώσουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τα προγράμματα που έχουν ε, κακές επιδόσεις. Τα προγράμματα που δεν δίνουν, ας πούμε, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ούτως ώστε στην έκθεση με τις αξιολογήσεις σας και στην τελική συμφωνία με το Συμβούλιο να βάλουμε, να λάβουμε υπόψη μας ε, αν χρειαστεί να κάνουμε τέλο πάντων περικοπές, πού να τις κάνουμε. Και για να λάβουμε υπόψη μας και εσά και τις απόψεις σας για το πού πρέπει να περικόψουμε ε, και πώς πρέπει να περικόψουμε. Ευχαριστώ. έδωσα, ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λαβία. Έχουμε μια διαδικασία, σωστή νομίζω. Έχουμε μαζέψει όλε τις προτάσεις πιλωτικών προγραμμάτων από την Επιτροπή και διαπιστώνω ότι ε, δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα δικό μου, αν και υπέβαλα τρία. Δεν ξέρω πού είναι, πρέπει να το δω, γιατί πριν από εβδομάδε τα υπέβαλα. Τέλο πάντων, θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο για το σχέδιο προπολογισμού. Έτσι κάναμε και πέρσι και τώρα έτσι θα κάνουμε. Αν περιμένουμε το Συμβούλιο θα πάμε στις διακοπές, στις ερηνές διακοπές, οπότε δεν θα προλάβουμε. Τα πιλωτικά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις τον Ιούλιο θα τα ψηφίσουμε και θα εξουσιοδοτήσουμε τον εισηγητή ε, τις προτάσεις να τις διατηρήσει για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού. Ε, είναι σωστό νομίζω αυτό. Έτσι κάναμε και την περασμένη φορά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Είναι το πιο σωστό. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε το Συμβούλιο γιατί μετά θα αργήσουμε πολύ. Ο κύριος Λόκεγκαρτ που είναι και ο συντάκτης της νομοδότησης Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Λαβία που ήρθε εδώ και μας ε, ενημέρωσε. Θα αναφερθώ σύντομα στη διαδικασία για να κατανοήσετε τι συμβαίνει όπως και εσύ, έχουμε πολλά κυρία δημοσιονομικά καθήκοντα, έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα, έχουμε ε, και τις νομοδοτήσεις για τις κυρίες προτεραιότητες. Ε, για το λόγο αυτό υπάρχει ένα πακέτο, ε, μια δέσμη ενημέρωσης που μοιράστηκε στους βουλευτές. Ελπίζω όλοι να λάβατε αυτή τη δέσμη των εγγράφων. Αν όχι, θα το λάβετε λέγεται ότι θα έχουμε τι γραμμές του προπολογισμού για τι οποίε εμεί έχουμε συγκεκριμένε ευθύνε ω Επιτροπή, έχουμε και χρονοδιάγραμμα, αναφέρονται για κάποιε προθεσμίε. και επίση έχουμε και το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον τύπο από την Επιτροπή και αναφέρονται εκεί κάποια από τα κυρία στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Ε, έχουμε το σχέδιο του προπολογισμού, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 25 Απριλίου. Και τώρα είναι η σειρά του Συμβουλίου να τοποθετηθεί όπως αναφέρθηκε και πέρσι η θέση του Συμβουλίου ήρθε πάρα πολύ αργά όπως είπε και η κυρία Πακ τέλη Ιουλίου προκειμένου να είναι αρκετά διαφανής η διαδικασία της κατάρτισης του προπολογισμού η δική μας Επιτροπή θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που ακολούθησε και πέρσι. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες του προπολογισμού ήδη τον Ιούλιο και όπως ήδη αναφέρθηκε θα μου δοθεί ελπίζω μια ζώδια εντολή ε, για να παρουσιάσω τις κατάλληλες τροπολογίες ε, για το Σεπτέμβριο και αν χρειαστεί για την αποκατάσταση του σχεδίου του προπολογισμού. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και αν θα χρειαστεί. Πρέπει να θέσουμε κάποιες ε, προτεραιότητες, όπως και πέρσι, καθώς δεν έχουμε πολλά περιθώρια, κυρίως ε, στον τομέα 3β, όπου έχουμε 25,6 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και το τομέα 1α, 91 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν και τα δύο αυτά νούμερα είναι κάπως πιο υψηλά από τα δύο τελευταία έτη. Προσπάθησα να δω ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω, ίσως λόγω της κατάστασης που έχουμε με τις πληρωμές. Παρ' όλα αυτά είναι θετικό που έχουμε 25,6 εκατομμύρια, καθώς πριν είχαμε μόνο 15. Παρ' όλα αυτά πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες ε, και ήδη ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, αλλά σε έρθω τώρα στα πιλωτικά προγράμματα. Ήδη είχαμε την προθεσμία, δεν ξέρω γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί το κείμενο της κυρίας Πακ, αλλά θα το δούμε και αυτό το θέμα και θα μάθουμε. Έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος και σας έχει διανεμηθεί. Είδα κάποιους να μοιράζουν αυτό το κατάλογο, νομίζω ότι το έχετε στη διάθεσή σας. Και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μέχρι τις Ιουνίου. Κατόπιν ε, η Κομισιόν θα εξετάσει αυτές τις προτάσεις και θα υπάρχει ένα feedback. Και έτσι λοιπόν θα δούμε τι είναι πλέον εφικτό όπως αναφερθήκε ήδη από το Γενικό Εισηγητή. Ήδη είχαμε την πρώτη συνάντηση με τους Κιώδης για να συζητήσουμε τις ε, προτάσεις ε, για τις δεσμεύσεις αναλήψης υποχρεώσεων και τις υποχρεώσεις πληρωμών, αλλά υπήρξε τουλάχιστον μία συνένεση να συνεχίσουμε με τις ε, συμπράξεις και με τον αθλητισμό που ήδη είχαμε υιοθετήσει πέρσι. Και κάποια λόγια για την γνωμοδότηση, για το προϋπολογισμό. Ε, η Επιτροπή υιοθετεί μια πρόταση για τις προτεραιότητες προϋπολογισμού για το 2013. Εγώ θα παρουσιάσω τον Ιούνιο το σχέδιο της γνωμοδότησης και θα ψηφίσουμε στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τώρα για τα προγράμματα διαβημάθηση και νεολαία σε δράση σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και εφαρμόζονταν πάντοτε, όπως και το πρόγραμμα Εράσμους. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα προγράμματα αυτά που δεν καλύπτεται. Έτσι λοιπόν πάντοτε για την μας ε, επιτροπή αποτελεί προτεραιότητα οι επενδύσεις ε, σε αυτούς τους τομείς και συνάδει αυτό και με τους στόχους του 2020. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης και να ε, επενδύσουμε σε δημιουργικούς τομείς και επίσης ε, πρέπει να έχουμε προτεραιότητες και στις ε, πολιτικές επικοινωνίας. Θα πρέπει να διαδίδουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό καθίσταται όλο ένα και πιο σημαντικό γιατί έχουμε και τις ευρωεκλογές του 2014. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα αυτά είναι τα κυρία σημεία για αυτές τις τρεις δράσεις που θα παρουσιάσουν στο μέλλον. Όμως ε, θα έχουμε και περισσότερες συνεδριάσεις ε, και θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανες, Ιβάν. Ευχαριστώ. Θα πω δύο λόγια για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα, αν και είναι πολύ καλά και καλύπτουν θέματα όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η... ο αθλητισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, δεν θα λάβουν ε, το σύνολο της χρηματοδότησης. Γνωρίζουμε και από τα περασμένα έτη και ακούσαμε και τι μας είπε και ο εισηγητής, ε, ότι μπορούμε να τοποποιήσουμε τον υπολογισμό. Στην Επιτροπή Προπολογισμών έχουμε κάποια επιρροή και νομίζω ότι οι προπαρασκευαστικέ δράσει, όσο αυτή για τον αθλητισμό, που σημείωσαν επιτυχία, θα πρέπει να συνεχίζει να χαίρει χρηματοδότηση. Ιδίω αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε ειδική χρηματοδότηση για τον αθλητισμό. Και θα ήθελα να πω στον συγγητή ότι ούτε η εκπαίδευση ούτε η νεολαία παρουσιάζονται ως προτεραιότητε στον προπολογισμό του 2013, ενώ στο παρελθόν εμφανίζονταν. Δεν ξέρω αν παρανόησα κάτι, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι το 2013 θα είναι η πιο δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του δημοσιονομικού, του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί ουσιαστικά ε, θα λειτουργήσουμε με όσα χρήματα μας έχουν απομείνει από τα περασμένα έτη. Φτάνουμε δηλαδή στα όρια τα δημοσιονομικά. Αλλά αν δούμε την ανεργία στους νέους και αν δούμε πόσο δυσκολεύονται οι άνθρωποι να προσαρμοστούν ε, στις νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Ε, νομίζω ότι η οικονομική κρίση μας έδειξε ότι χρήζουν βοήθεια οι νέοι και θα πρέπει να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί θα επαναληφθώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σιγητή για την εξαιρετική δουλειά του και την εξαιρετική παρουσίαση. Θα είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Για τη δική μας ομάδα είναι προφανεί ε, οι προτεραιότητε. Η διαβίου μάθηση έρχεται σε πρώτη θέση, όπως ε, και στα προηγούμενα οικονομικά έτη. Εδώ βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε τις ε, δεσμεύσεις ανάπτυξης υποχρεώσεων και τις πιστός πληρωμών για τη διαβίου μάθηση. Και ελπίζω ότι και στο ε, μέλλον η διαβίου μάθηση θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα ξεκινώντας από το 2013 και έχουμε και την γραμμή 3 3Δ, ε, το πρόγραμμα για τα ΜΜΕ, για τους πολίτες, για την ηθαγένεια και θα θέλαμε να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο οι δεσμεύσεις ε, Άκουσα τι είπε ο κύριος Λαβίου, από το 2013 θα πρέπει να είναι σαφή τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά αυτές τις προτεραιότητες. Ε, θα πρέπει ε, να παραμείνουν ως έχουν με ορίζοντα το 2020. Θα πρέπει φυσικά να επιμείνουμε εκεί, ξεκινώντας από το 2014. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι υπάρχει ευρεία συνένεση για τον αθλητισμό κατατέθηκαν πολλές προτάσεις για προπαρασκευαστικές δράσεις, συγκεκριμένα για το τρέχον έτος. Ε, είμαστε στα 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι και πάρα πολλά. Ε, αυτά τα χρήματα θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης ε, για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα στον τομέα του αθλητισμού και θέλω να αναφέρθω και στο έγγραφο εργασία με τι προτεραιότητε για τι προπαρασκευαστικέ δράσει για τα επόμενα έτη. Θα χρειαστεί να τα διατηρήσουμε αυτό στο πλαίσιο του προπολογισμού έτσι λοιπόν ε, έχουμε την καταπολέμηση ε, του κοινωνικού αποκλεισμού των μειονεκτουσών ομάδων. Ε, πρέπει επίσης να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη και την προώθηση των σωματικών δραστηριοτήτων για να βελτιώσουμε τη δημόσια υγεία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που εγώ χαιρετίζω. Και να μιλήσω αγγλικά. κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, μαζί με την κυρία Γκέντση και την κυρία Σιλβία Κώστα ε, θα επικεντρωθούμε στο θέμα της πρόσβασης του Πανεπιστημίου για τους νέους ε, Ρωμά. Υπάρχει μια σχετική πρόταση την περασμένη εβδομάδα, συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο και συζητήσαμε περίπου 20 προτάσεις θα πρέπει φυσικά να περιμένουμε και την απόφαση της Κομισιόν, ε, αλλά ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θα ψηφίσουμε προς την κατεύθυνση που προτείνει και ο συγγετής. Νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική βάση. Ίσως θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ε, ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι πολύ ποιοτική. Μάλιστα, πολύ σύντομα, γιατί ο συνάδελφο, ο κ. Λεβί από την Επιτροπή Προπολισμού ε, παρευρίσκεται εδώ. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, ήδη συζητούνται δυνατότητες ε, περικοπών, εξοικονομήσεων, πόρων για κάποιες δράσεις όπου δεν είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Όμως νομίζω ότι το δική μας Επιτροπή έχει πάρα πολύ μικρό προπολογισμό και έχουμε καλά ποσοστά εφαρμογής. Και φυσικά έχουμε και ιστορίες επιτυχίας να αφηγηθούμε. Ε, γιατί πράττουμε καλά πράγματα υπέρ των Ευρωπαϊκών πολιτών. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να παρουσιάσω εγώ εδώ, ότι εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα περικοπών για το δικό μας προπολογισμό, γιατί πρέπει να προωθήσουμε τους τομείς της εκπαίδευσης, αυτών των δραστηριοτήτων όπου συμμετέχουν οι νέοι, οι πολίτες, να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που πρέπει να βγει από την Επιτροπή μας. Την τροπολογία μου την είδα. Έκανα κι εγώ κάποιες τροπολογίες στον πολιτισμό θα τις είδατε κι εσείς. Είναι από καιρό. Δεν ξέρω που μπερδευτήκαμε. Όχι από το γραφείο μου γιατί συνήθως είναι πολύ προσεκτική. Μόνο έτσι μπορούμε να εργαστούμε, όπως είπα και γρήγορα, με τα αγγλικά. Να συμφωνήσουμε, να δουλέψουμε στα αγγλικά. Ας το δεχτούμε αυτό για να προλάβουμε και να μην περιμένουμε το Συμβούλιο. Οπότε ζητώ τη σύμφωνη γνώμη σας ότι θα προχωρήσουμε έτσι. Και ποιος κυρίως από την Κομισιόν. Α, η κυρία Μπριζίτ. Κυρία είναι. κυρία Μπριζίτ Εγκός. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν είναι εδώ ο κύριος Νότ. Μας γενικά σχόλιο και για να επαναλάβω σε υπόθηκαν η παιδιά και ο πολιτισμός ε, έλαβαν ε, ε, πρόσθετες, πρόσθετα κονδύλια για να προωθηθεί η απασχόληση σύμφωνα με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 για το πρόγραμμα της διαβίωμασης. Είχαμε 13,6 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι είχαμε στο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα και για το πρόγραμμα νεολαία δράση περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 13 εκατομμύρια παραπάνω από την αρχική πρόβλεψη. Και αυτό τονίζει το πόση σημασία δίνει η Κομισιόν σε αυτά τα δύο προγράμματα. Για τα υπόλοιπα προγράμματα Δυστυχώ ε, έπρεπε να ακολουθήσουμε το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, δηλαδή ήταν ε, πολύ μικρές ευξήσεις για τον πολιτισμό και για τα μέσα ενημέρωσης, ε, ήταν λίγο παραπάνω από 1%. Για τον αθλητισμό θα καλωσορίζουμε οποιαδήποτε προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα. Και τα περιθώρια ήταν αρκετά στενά και η Κομισιόν προσπάθησε να σεβαστεί ε, αυτά τα περιθώρια και στο τίτλο 1α και 3β. Και έτσι εξηγείται γιατί δεν λαμβάνουμε παραπάνω χρηματοδότηση. Παραπάνω κονδυλίσεως να δώσω το λόγο και στο συνάδελφο που είναι υπεύθυνο ε, για τον τομέα της ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Να πω ότι ο προπολογισμό για την επικοινωνία συνεχίζεται χωρίς μεγάλες αλλαγές ε, και έχουμε ήδη κάτι θετικό στο σημερινό πλαίσιο. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες, μόλις λάβουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό, γιατί θα θέλαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο ταχείς στο να εξετάσουμε όλες τις προτάσεις ε, τροπολογιών σε σχέση με πέρσι. Γιατί ε, εξακολουθούμε να έχουμε ε, κάποιες επιφυλάξεις ε, για τον περσινό προπολογισμό. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια καλύτερη κατάσταση φέτος, να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα γρηγορότερα. Έτσι λοιπόν θέλω να λάβουμε τις πληροφορίες το συντομότερο και θα συζητήσουμε μαζί σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να λύσουμε εκ των προτέρων δυνατόν τέτοιου είδους προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο, κύριε Λαβία. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη χρήσιμη συζήτηση. Νομίζω ότι προκύπτει κάτι ξεκάθαρα αφενός ε, των ενδιαφέρον της Επιτροπής για προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα αφετέρου το ότι στους τομείς όπου θα ενταχθούν περισσότερες προτάσεις ότι υπάρχουν πολύ συγκρατημένα περιθώρια και είναι σαφές ότι αυτό θα μας σωθήσει στο να χρησιμοποιήσουμε τις προτεραιότητες που θα καθορίσει αυτή η Επιτροπή έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα το περιθώριο που έχουμε. Και θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο Ιβάν ο οποίος δεν ε, μπόρεσε να βρει την αναφορά της υποστήριξης στους νέους και στην κατάρτιση των νέων. Καταρχήν, μεταξύ των προτεραιοτήτων του προπολογισμού του 2013, από την αρχή της διαδικασίας θέσαμε ε, ως προτεραιότητα τους νέους ε, και την απασχόληση των νέων. Ήταν μεταξύ των ε, κυρίων προτεραιοτήτων του προπολογισμού, αλλά και στο στερικό της εντολής για τον τρομερή διάλογο που προετοιμάζουμε και που θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο, στο σημείο 44, τα προγράμματα ε, πολιτισμού και παιδείας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι ε, είναι δύσκολο στη συνέχεια να αναφέρουμε όλε τι γραμμέ προπολογισμού. Λέμε από την αρχή ότι έχουμε κάποια προγράμματα που είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όπως το διαβίου μάθηση, το νεολαία σε δράση κτλ. Και σίγουρα πρέπει να υποστηριχτούν στο Κοινοβούλιο και φυσικά θα δοθεί και κατάλληλη υποστήριξη από εμά. Okay, thank you very much. dass Sie hier waren, lieber Herr Kollege Damit schließen wir den Punkt. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε το σημείο 12 στα γρήγορα το 13 για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλετε τώρα να πείτε κάτι, τα είπαμε όλα. Έλεγα ότι προχωρούμε στο σημείο 13. I have no further comments on no. Δεν έχω άλλα σχόλια για το 13. Έχω για το MFF, το πολιτές δημοσιο... Ε, α, για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Α, όχι τον προϋπολογισμό για το 2020, το πολιετές, στο σημείο 13. Όχι για τον προϋπολογισμό του 2013, για το πολιετές, στο σημείο 13. Για την περίοδο 2014-2020. Θα είμαι σύντομος. Η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού που γίνεται στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, MFF, για λόγους συντομίας, μέχρι σύντομα το MFF ήταν διοργανική συμφωνία. Πολιτική συμφωνία παρά νομοθετικό κείμενο, κείμενο νομοθετικού περιεχομένου από την άλλη πλευρά. Το MFF θεσπίζει τον πολιετή προϋπολογισμό και τα πολιετή προγράμματα. Ε, η συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε το καθεστώς του MFF και τώρα είναι κανονισμός, στηρίζεται σε κανονισμό του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πει ναι ή όχι, χωρίς να αλλάζει την πρόταση. Το τωρινό τελειώνει τέλος του 2013, το δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF το τωρινό. Στην προσωρινή Επιτροπή του Κοινοβουλίου αναφέρονται οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου για το νέο MFF και η Κομισιόν τον περασμένο Ιούλιο έκανε προτάσεις και τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τον ίδιο τον κανονισμό. Η διαδικασία σύμφωνης γνώμης είναι συγκεκριμένη και προβλέπει ε, διάμεση έκθεση. Αυτή θα είναι έκθεση μη νομοθετική, αλλά παρουσιάζει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για το επόμενο MFF. Η Επιτροπή Προπολογισμού τον Οκτώβριο θα αποφασίσει, όλες οι επιτροπές θα υποβάλουν γνωμοδοτήσεις. Εγώ τον Ιούλιο ε, υπέβαλα ένα σχέδιο γνωμοδότησης, ε, θα υποβάλω σχέδιο γνωμοδότησης και θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό το τι θα πούμε στις νομοδοτήσεις μας, γιατί πάνω εκεί θα στηριχθεί η Επιτροπή Προϋπολογισμού για να συμπεριλάβει ως προτεραιότητες τα προγράμματά μας στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εγώ θα στηρίξω την γνωμοδότησή μου στα επιχειρήματα που αναφέρονται ε, ήδη ε, τα νούμερα ε, θα ακολουθήσω με τα, τις προτάσεις για το Εράσμους το και τα άλλα δύο προγράμματα. Ε, βέβαια με ενδιαφέρει να δούμε τι θα πούν και οι συνάδελφοι σε όλα αυτά. Yeah. Who wants the floor? Ποιος ζητάει το λόγο? Κανείς? Καλώς. Καλώς. Θα περιμένουμε το σχέδιο έκθεσης. Τότε θα συζητήσουμε. Τελειώσαμε και το 13. να ρωτήσουμε την Κομισιόν αν θέλει να παρέμβει. Θέλει. Γιατί σήμερα το πρωί θα, σας θέλαμε να μας πείτε κάτι, αλλά δεν είσαστε παρόντες. Τώρα είσαστε. Έλεγα ότι πάντα είμαι εδώ όταν με χρειάζονται, κυρία, όταν χρειάζομαι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. 100% αλήθεια. Απλώς ρώτησα αν θέλει κανείς να πει κάτι για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν ζητεί το λόγο κανείς, θα το συζητήσω μετατικά όταν θα υποβληθεί και το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τώρα θα πάμε στο σημείο 11. Πάμε πίσω. Εδώ το θέμα μας... Είναι η Ευρώπη για τους πολίτες. Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες είναι το θέμα μας εδώ. Και ο εισηγητής μας είναι ο συνάδελφος Χάνου Τάκουλα. Όπως ξέρουμε, εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το πρόγραμμα που το συζητήσαμε και με τους συντονιστές σήμερα. Δηλαδή, το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται σε μια πρόταση επί της οποίας θα πούμε ή ναι ή όχι. Το συζητήσαμε επί μακρόν σήμερα το πρόβλημα αυτό και καταλήξαμε ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας το θέμα δεν ρυθμίστηκε καλά για μας και δεν επιτρέπεται σε μία έκθεση για τους πολίτες εμείς να μην έχουμε καθόλου λόγο. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφαίνεται επί του και να καταθέτει τροπολογίες, εμείς όχι. Και είπαμε σήμερα το πρωί ότι θεωρούμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται, μας γελιοποιεί και πρέπει οπωσδήποτε να αντιταχθούμε. Η πρόταση που προέκυψε είναι να κάνουμε μια ενδιάμεση έκθεση όπως και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά βέβαια αυτά είναι στα στα μάτια το Συμβούλιο δεν υπόσχεται ότι θα μας λάβει υπόψη, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι πραγματικά γελίο. Το συζητήσαμε στους συντονιστές και εγώ πρότεινα να γυρίσουμε όλοι στις πολιτικές μας ομάδες και από εκεί να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε πλειοψηφία για την απόρριψη της πρόθεσης θα την απορρίψουμε και αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τίποτε. Δεν θα έχουμε κανένα πρόγραμμα. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν εν τη αυτή περιπτώσει τι θα κάνουν. Διότι πρώτον πρέπει να δαπανηθούν τα υπάρχοντα κονδύλια και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Είμαστε ένα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογέ και δεν επιτρέπεται να μην έχουμε πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Αλλά ούτε έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες χωρίς να έχουμε συμμετάσχει εμείς. Αυτή ήταν η άποψη που διαμόρφωσαν οι συντονιστές. Είπαμε ότι θα πάμε στις πολιτικές μας ομάδες και θα το συζητήσουμε εκεί το θέμα. Αν συμφωνήσουν οι πολιτικές ομάδες ότι θα το αφήσουμε αυτό το θέμα, δεν θα το επιχειρήσουμε, θα πούμε όχι, θα το απορρίψουμε. Και εκείνοι που έχουν άλλη άποψη από τη δική μας νομική υπηρεσία πρέπει να έρθουν και να μας ε, το εξηγήσουν. Γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα με βάση τη νομική μας υπηρεσία. Σας είπα τα σχετικά με τους συντονιστές και δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή που περιμένει, ο Χάνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι μπορώ να προσθέσω τώρα. Όπως το συνοψίσατε, ήταν σωστό. Ε, αυτή ήταν η συζήτηση που διεξήχθη. Όλοι είμαστε έκπληκτοι από το αποτέλεσμα. Τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν δεν αρέσκονται στην ιδέα του να υπάρχουν δύο ενότητες. Η καλύτερη λύση θα ήταν να αποφασίσουν οι πολιτικές ομάδες. Γιατί σε κάποιο βαθμό θα αποτελέσει προηγούμενο για το πώς θα λειτουργεί η συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου, θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Αλλά τελικά έχει δίκιο η Πρόεδρος. Ας πάμε στις πολιτικές ομάδες και ας δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα αυτό, πολύ καλό πρόγραμμα επίσης και τι θα πρέπει να γελιοποιηθούμε. σε μια δημοκρατία η ψήφος δεν έχει την έννοια της επικύρωσης ή της απόρριψης μόνο. Ας δούμε λοιπόν αν μπορούμε να συντάξουμε αυτά τα δεδομένα μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ η Κομισιόν. Θέλει να πει κάτι. Με την κυρία Ρέντινγκ μιλήσαμε πολύ και με την νομική υπηρεσία της Κομισιόν Ξέρουμε τη γνώμη της κυρίας Ρέντινγκ. Ακούσατε ότι αποφασίσαμε να σκληρύνουμε τη στάση μας όμως και να μην ακολουθήσουμε αυτόν τον ρεαλιστικό δρόμο σε εισαγωγικά μιας εικονικής συναπόφασης όπως πρότεινε η κυρία Ρέντινγκ στην τελευταία συνεδρίαση. Θέλετε να πάρετε θέση πάνω σε αυτό, παρακαλώ. Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω τις ανησυχίες σας, τις καταλαβαίνω. Είναι ένα θέμα που ξεπερνάει αυτό το πρόγραμμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το άρθρο 352 δεν ήταν όμως η καλύτερη επιλογή κατά την Κομισιόν άρθρου. Αναλύσαμε όλες τις δυνατότητε. θα προτιμούσαμε το Κοινοβούλιο να είναι συνομοθέτης. Ζητήσαμε και πλήρη νομική ανάλυση από τις νομικές μας υπηρεσίες και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Και η μόνη λύση ήταν να βασιστούμε τελικά στο άρθρο 352. Να σας υπενθυμίσω, συνάδελφοι, ευρωβουλευτές, για τους ευρωβουλευτές που δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση με την κυρία Ρέντινγκ, δηλαδή, ότι η ουσία του προγράμματος είναι το βασικό. Το κέντρο βάρους του προγράμματος ε, βρίσκεται στη δημοκρατική συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή. Αυτό είναι το βασικό στατικό του προγράμματος. Φυσικά υπάρχει και το θέμα της μνήμης αυτό θα μπορούσε, θα να έχει συνδεθεί με το 1,67. Αλλά αυτό είναι δευτερεύουσα σχέση με την συμμετοχή. Μέσω της μνήμης ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την αίσθηση των Ευρωπαίων πολίτων ότι ανήκουν κάπου. Μην το ξεχνάτε λοιπόν αυτό. Αυτή η αλλαγή προσέγγισης συνάδει και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και με τα νέα άρθρα 10 και 11, όπου η συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ένα στόχος που αναφέρεται ρητά συνθήκες, στη συνθήκη. Αλλά τα άρθρα αυτά δεν μας δίνουν την εξουσία να εφαρμόσουμε προγράμματα. Γι' αυτό χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε το 352. Υπάρχει αυτή η μερική γενική συμφωνία στο μεταξύ του Συμβουλίου και η Προεδρεύουσα που ήταν και πρόεδρος εκείνης της συνάντησης είναι μαζί μας εδώ και μπορεί ίσως να προσθέσει κάτι σε αυτά που σας είπα εγώ. Στο Συμβούλιο, στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, η καθοριστική ε, σημασία της συμμετοχής, του participation, τονίστηκε ακόμα περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία. Η Κομισιόν χρειάστηκε να βασιστεί, να βασιστεί την πρότασή της στο 352. Αναγκάστηκε να το κάνει. Λόγω της νομοθετικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή διτή νομική βάση όταν ε, υπάρχει ασυμβατότητα των δύο νομικών βάσεων. Ο μηχανισμός με τον οποίο επιδρούν ε, στο 352 και το 167 ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι ασύμβατος μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισορροπία που προβλέπει η συνθήκη. Έχουμε ήδη ανταλλάξει επιχειρήματα, οι αρμόδιες δηλαδή νομικές υπηρεσίες, ξέρουμε το διακύβευμα, θέλουμε να ενισχύσουμε το επιχείρημα ότι μόνο μετά από ενδελεχή νομική ανάλυση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βασιστούμε στο άρθρο 352. Δηλαδή πραγματικά κάναμε νομική ανάλυση και μετά φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Και εμεί συζητήσαμε διεξοδικά και καταλήξαμε αλλού. Και εμεί έχουμε νομική υπηρεσία που λέει τα αντίθετα από αυτά που λέει η δικιά σα νομική υπηρεσία. Μα επιτρέπεται και είναι θεμητό να καταλήξουμε σε διαφορετικό συμπέρασμα και να πορευτούμε ανάλογα. Ε, και έχουμε και τον ε, ε κύριο Λένε και τη Νομική Επιτροπή που συμφωνεί με τη νομική μας υπηρεσία. Ε, τι περισσότερο να ζητήσουμε και να κάνουμε. Ε, φαντάζομαι ότι δεν σας ανησυχεί αυτό. Μπορεί όμως και λίγο να σας ανησυχεί. Ε, το Συμβούλιο θέλει να πει κάτι. Επιθυμεί να λάβει το λόγο το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την καταστροφή που έκανα. Λυπάμαι που ακούω το συμπερασμά σας. την απόφασή σα και θέλω να προσθέσω ότι αναμφισβήτητα μία από τις κύριε προκλήσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης της πρότασης ήταν η προτινόμενη νομική βάση που απαιτεί ομοφωνία του Συμβουλίου. Δεν ε, έχουμε τακτική νομική διαδικασία και θα έχουμε και σε ορισμένα κράτη-μέλη δύσκολε διαδικασίε λήψη αποφάσεων. Και Γι' αυτό το λόγο, κατόπιν αιτήματο των κρατών μελών, η Προεδρία αποφάσισε να ζητήσει γραπτή γνωματότηση της νομικής υπηρεσία. Να καθεσυχάσω την Επιτροπή και σας, Πρόεδρε, ότι το θέμα της νομικής βάσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο για το Συμβούλιο και ακούστηκαν πάρα πολλές ανησυχίες από τα κράτη-μέλη και σε σχέση με τον ειδικό ρόλο που δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα πω τώρα σε νομοτεχνικά ζητήματα γιατί δεν είμαι νομομαθής, αλλά καθώς το Συμβούλιο πιστεύει ότι έχουμε αυτές τις δύο θεματικές, ε, δεν είχαμε καμία επιλογή σε σχέση με την νομική βάση. Και θέλω να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σιγητή, τον κύριο Τάκουλα, για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ των ε, τριών εκπροσώπων ε, των νομικών υπηρεσιών στις 21 Απριλίου. Και όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς δεν κατέληξε η συνάντηση αυτή σε κάποια εξέβρεση λύσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράγματι, όταν ρωτάς ε, τρεις νομικούς, έχεις τρεις διαφορετικές γνώμες. Το ίδιο ισχύει για τις νομικές υπηρεσίες, από ό,τι φαίνεται. Ε, ε η δική μας νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν είναι τέτοια. να σχολιάσω κάτι που είπε η εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πρόκειται για δημοκρατική δέσμευση και συμμετοχή. Αυτό ήταν το πρόγραμμα και εμάς μας ενδιαφέρει η δημοκρατική δέσμευση και η συμμετοχή, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα αυτό. Γι' αυτό θυμώνουμε τόσο πολύ. Όλα καλά για τους πολίτες, αλλά και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών πρέπει να ερωτώνται αυτό έχει να κάνει με τη δημοκρατική νομιμοποίηση όλου του θέματος. Το Συμβούλιο εργάστηκε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα θαυμάσια και έκανε καλά πράγματα προσθέτοντας, αφαιρώντας. Θέλουμε και εμείς όμως να κάνουμε αυτό. Ο Χάνου Τάκουλα είναι εισηγητής και θέλει να υποβάλει καινούργιες ιδέες. Θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα που θεωρεί ότι δεν είναι σωστά στο πρόγραμμα. Δεν νομίζω για παράδειγμα ότι εγώ και τα σπίτια της Ευρώπης δεν θα τα χρηματοδοτούμε θα ε, καταστραφούν χρόνια δουλειάς. Εσείς δεν ε, κάνατε την ε, σχετική τρόπο πρόταση για αλλαγή στο Συμβούλιο. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Τον κοινοβουλευτισμό εγώ δεν τον ερμηνεύω έτσι, ούτε κανείς άλλος από τους παρευρισκομένους. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουμε πιο σκληρή στάση και θα καλέσουμε τις πολιτικές ομάδες να μας υποστηρίξουν που θα πούμε όχι και ο συνάδελφος ε, ε, λένε είναι της ίδιας άποψης. Και ας σκεφτούν η Κομισιόν και το Συμβούλιο μήπως θα πρέπει να κλείνουν προς την άποψη της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει η υπόθεση, διότι πλησιάζει το 2014 και πρόκειται για την δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Αλλά αν δεν έχουμε ε, συμμετάσχει και εμείς, δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατική συμμετοχή. Ε, στο, για πρώτη φορά έχουμε διερμηνία στα κροατικά, στην καμπίνα υπαριθμών 27. Ε, είναι πολύ ευχάριστο που μπορείτε να παρακολουθείτε τη μητρική σας γλώσσα, αν και ξέρω ότι καταλαβαίνετε καλά και τα γερμανικά και τα αγγλικά. Ε, χάνουν, τα είπαμε όλα, μήνε, γιατί ακόμα σε χρειαζόμαστε. Κλείνει η συζήτηση. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την παρουσία της. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο για την παρουσία του. Και επανέρχομαι σε ένα θέμα που αναφέραμε. Πού είναι ο κύριος Λόκεγκάρντ. Έφυγε. Στην συνεδρία των συντονιστών είπαμε ότι οι συντονιστές και εμείς θα αποφασίσουμε για τη γραμμή του προϋπολογισμού για αυτό το αποθεματικό, να το καταργήσουμε. Η Κομισιόν υποσχέθηκε ότι εργάζεται πάνω στο θέμα Μίλησε και με τον κύριο Φόλκερ και θεωρεί ότι μέχρι μέσα Ιουνίου έχει χρόνο, όπως και ο κύριος Λόκεγκαρντ, αλλά νομίζω ότι το χρονικό ορίζοντα δεν τον είχαν αντιληφθεί σωστά. Τώρα, έστειλε ένα σχέδιο σήμερα το μεσημέρι και τονίζει ότι είναι σχέδιο. Γι' αυτό δεν θα διανεμηθεί σε όλους. Δεν το είδε κανείς εκτός από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Το έδωσε στον κύριο Λόκεγκαρτ με την παράκληση να το δει. Το είδα και εγώ και η κυρία Τρούπελ επίσης. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι έκανε κάποιες σκέψεις η Κομισιόν προς τη σωστή πιστεύω κατεύθυνση, ε, στρατηγικές κατευθύνσεις, ανάδυση νέας πραγματικότητας, νέες λέξεις χρειάζονται, το περιβάλλον αλλάζει γρήγορα με επιπτώσεις, η πραγματικότητα εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ. Α, προς τη σωστή κατεύθυνση πάει, νομίζω ε, ε, έτσι είναι το σωστό η επικοινωνία εξελίσσεται, συνδυάζουμε τις δυνάμεις στην επικοινωνία, σταθερότητα, αλληλεγγύη, ανάπτυξη κτλ. κτλ. Ή θυμίζομαι τον απότερο σκοπό της Ένωσης. Τέτοια θέλουμε από την Κομισιόν να μας λέει. Ε, ε, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση λοιπόν αν τα αντιλαμβάνουμε τα πράγματα σωστά. Είναι μια συλλογή ιδεών αυτό το σχέδιο και μέχρι μέσα Ιουνίου θα είχαν ολοκληρώσει την άποψή τους. Τώρα, μια θερμή παράκληση. Ο κύριος ε, Φόλκερ θα μπει σε λεπτομέρειες, θα κάνει πιο εκλεπτισμένο το κείμενο, θα πάρει και ένα κείμενο από τον κύριο ε, Φόλκεγκαρντ για να το κάνει καλύτερο, τον κύριο Λόκεγκαρ, συγγνώμη, και η Επιτροπή Προϋπολογισμών αύριο ή μεθαύριο που θα συνεδριάσει θα αποφασίσει να ε, άρει αυτό το, από το απόθεμα. Δεν ξέρω την φίβρα, αλλά τέλο πάντων είναι σωστό τώρα το εξή. Έχουμε το πρώτο σχέδιο σε αυτό το κείμενο που εργάζεται ο συνάδελφο και χαίρομαι που λάβαμε τόσο γρήγορα αυτό το σχέδιο κειμένου καθώ πρέπει να λάβουμε και μία απόφαση. Δεν έχω αμφιβολία ότι η ομάδα εργάζεται σκληρά για να μας παρουσιάσει κάτι χρήσιμο και μπορώ να πω ότι έχουμε μια καλή συνεννόηση για το τι πρέπει να πετύχουμε. Η μόνη μου ανησυχία είναι ότι μήπω ε, λαμβάνοντα αυτή την απόφαση τώρα διακόπτουμε αυτή την ευαίσθητη διαδικασία. Και όπως είπα ήδη επανειλημμένο σήμερα, για μένα δεν είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε τώρα. Έκανα μια έρευνα σήμερα το απόγευμα για το θέμα αυτό και φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα να το αναβάλουμε για δύο-τρεις εβδομάδες. Στις 19 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Προπολογισμών ε, και οι συνάδελφοι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να λυθεί και η απόφαση και εμείς συνεδριάζουμε στις 19 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν ε, είναι πρακτικό το ζήτημα πρακτική οργάνωση να το εξετάσουμε αυτό το θέμα, να το διεκπαιρεώσουμε και να συνεργαστούμε και να μην ε, αγχωθούμε. Και όπως είπατε, θα συμφωνήσει και με τον κύριο Πολκό. Και οι δύο συμμετέχουμε σε αυτό. Δεν έχουμε βέβαια φτάσει ακόμη στη συμφωνία και φαίνεται να μην ε, είναι σκόπιμο να λάβουμε αυτή την απόφαση τώρα, γιατί έχουμε την ευκαιρία να περιμένουμε μέχρι τις 19 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν, ε, απευθύνω έκκληση να λάβετε αυτή την απόφαση επίσημα να αναβληθεί αυτή η διαδικασία λέγοντας όχι τώρα, μόνο και μόνο για να έχουμε χώρο και χρόνο να ολοκληρώσουμε αυτήν την καλή δουλειά που κάνουμε από κοινού. Δηλαδή είμαστε στο ίδιο σημείο που είμαστε σήμερα το πρωί. Εμένα μου είπαν ότι αν δεν μπούμε ναι ή όχι τώρα, αύριο ή μεθαύριο η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα το δεχτεί και μετά δεν, θα πούμε τίποτα άλλο. Θα αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα. Πρέπει να πούμε τώρα όχι. Για να πούμε κάποια στιγμή το ναι στο μέλλον. Αλλά είναι λίγο αστείο αυτό το πράγμα. Δεν χρειαζόταν να κάνω όλη αυτή την προσπάθεια να κινητοποιήσω τον κύριο Φόλκερ και να του πω να μας δώσει αυτό το ατελές κείμενο. Ε, εγώ είχα μια συγκεκριμένη εντύπωση ότι θα ε, συμφωνούσαμε και μέχρι τις 15-17 θα είχε το έτοιμο κείμενο. Θα έπρεπε να, και μάλιστα σε πολλά σημεία είναι πιο αυστηρό το, αυστηρή η πρότασή του από αυτή που έχουμε τώρα. Πώ είναι δυνατόν να πιέζουμε κάποιον ο οποίο είναι καλοπροαίρετο. Ο κυρίος Βόλκερ είναι ένα καλό μα συνεργάτη ε, ανέλαβε το αξίωμα του αργότερα, αλλά έχει καταλάβει ε, περί τίνος πρόκειται. Ε, δεν ε, έχει ε, τη δυνατότητα να δράσει μόνος του όμως, έπρεπε να κάνει πολλές διαβουλεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την Επίτροπο Ρέντινγκ, δεν μπορεί μέσα σε τρεις μέρες και του είπαμε μέχρι τις 17. Τώρα να τρέπονται αυτά τα προγράμματα. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την απόφαση που λάβαμε σήμερα. Ο κύριος Λόκεγκαρ πάλι και μετά θα ρωτήσω και τη γνώμη των συναδέλφων. Εγώ δεν είμαι βέβαια απαντογνώστης εδώ, θα ακούσω τη γνώμη σας. Ο κύριος Λόκεγκαρτ πάλι. Κατανοώ ότι πρέπει να το επιλύσουμε αυτό το θέμα. Αλλά δεν ξέρω πού να εξυπηρετούμε αν το κάνουμε τώρα. Δηλαδή και εμείς ε, και η Κομισιόν και η Επιτροπή Προπολογισμών θα είναι πλήρως ικανοποιημένοι με, με συμφωνία στα μέσα Ιουνίου. Γιατί λοιπόν, για ποιον το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα ως Επιτροπή, ως Κοινοβούλιο, αν έχουμε στη διάθεσή μας δύο-τρεις εβδομάδες παραπάνω για να διαπραγματευτούμε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτό το επιχείρημα με πάνω σεβασμό δεν φαίνεται ότι διαφωνεί κανεί ότι καλό θα ήταν να έχουμε δύο-τρει εβδομάδε ακόμη. Δεν καταλαβαίνω ποιον ενοχλούμε αν κάνουμε κάτι τέτοιο, εκτό ίσω από την Κομισιόν. Αλλά 6-9 μήνε προσπαθήσαμε και αγωνιστήκαμε να έρθουμε σε αυτό το σημείο και τώρα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε κάτι και θα χρειαστούμε απλώ δύο-τρει εβδομάδε ακόμη. Αυτή είναι η κοινή συνεννόηση μεταξύ ημών και Κομισιόν δεν καταλαβαίνω γιατί όχι λοιπόν. Πήραμε διαφορετικέ οδηγίε. Εγώ ρώτησα τη γραμματεία της Επιτροπής και μου είπανε ότι έπρεπε να αποφασίσουμε σήμερα και ότι στις 7 Ιουνίου, όχι, όχι αύριο 31 θα αποφάσιζαν και αν δεν πούμε τίποτε θα περάσει ή θα λέγαμε εμείς όχι, θα πούμε όχι, οπότε το αναβάλουμε για την ημέρα του Αγίου ποτέ. Ή θα περιμένουμε τον κύριο Φόλκερτ να μας ολοκληρώσει αυτό που άρχισε. Ε, Μάρκος Κουρία, τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε όχι και να περιμένουμε ή να πούμε ναι. Μάρκος Κουρία. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση εδώ, γιατί έχουμε διαφορετική ενημέρωση, αν ακούσω ότι είπε ο κύριος Λόκεκαρτ και όσοι είπε η να πουμε ναι μαρκος κουρια πιστευω οτι υπαρχει καποια συγχυση εδω γιατι εχουμε διαφορετικη ενημερωση αν ακουσω οτι ειπε ο κυριος λογκεκαρτ και οσο ειπε η κυρια Πακ αν ε, ε, τα πράγματα είναι όσο έχει, όσο ε, λέει η κυρία Πακ, νομίζω ότι ούτε πρέπει να χάσουμε χρόνο, ούτε να πούμε όχι για να επανέλθουμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, αν πρέπει μέχρι μεθαύριο, μέχρι αύριο να δώσουμε την απάντησή μας, δεν μπορεί να είναι θετική. Συμφωνώ με τον Μάρκο Κουρία αν έχουμε χρονική πίεση και έτσι κατάλαβα και την Χέλγα Τρούπελ ότι αύριο θα ε, αποφασίσουν στους προϋπολογισμούς. Ε, α, μεθαύριο, καλά. Μεθαύριο. Τότε θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κύριο Φόλκερ ότι περιμένουμε να υποβάλει το κείμενο όπως συνεννοηθήκαμε και όπως συνεννοηθήκατε κι εσείς μαζί του. Να το διατυπώσει και να το δώσει. Θα είναι αυτό ε, ένα κείμενο που θα στηρίζεται στην εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Σε αντίθεση της περίπτωση μπορούμε να προβλέψουμε ένα άλλο αποθεματικό. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να τον μπλοκάρουμε γιατί υπάρχουν ορισμένα ε, πράγματα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το αποθεματικό. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε σαφές μήνυμα στον κύριο Φόλκερ. Λοιπόν, ε, η Χέλγα. Εγώ σήμερα το πρωί προσπάθησα να συνεννοηθώ και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις επιθυμίες του κυρίου Λόκεγκαρτ, για να καταλήξουμε σε μια πρόταση σχετικά με το τι θα κάνουμε. Ε, μας είπες πόσο κατεπήγον είναι και, έχουμε και τον κύριο Φόλκερ, ο οποίος ε, κάνει μια προσπάθεια για λογαριασμό μας. Δεν είμαι η συντονίστρια για τους πρασίνους, αλλά μπορώ να συμφωνήσω ε, νομίζω με την ε, κυρία Κάμερεφερτ Μικρόφωνο. Λοιπόν, θα με θετικό μήνυμα στον κύριο, στο, στην Επιτροπή Προβλήσεων. Θα στείλω μία ε, κατεπίγουσα επιστολή, πολύ ευγενική στον κύριο Φόλκερο, ότι ε, θα άρουμε το αποθεματικό ε, δείχνοντας μια εμπιστοσύνη αλλά ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθεί στις επιθυμίες μας και τα αιτήματά μας και θα μας δώσει το κείμενο μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Είναι καλό αυτό? Εντάξει. Τελειώνουμε λοιπόν τη συζήτηση και πάμε στο σημείο 14. Ναι, κύριος Λόκεγκάρτ. οι βουλευτέ προσπάθησαν να το παρουσιάσουν αυτό με κατάσταση που χρειαζόμαστε περισσότερη εμπιστοσύνη. Εκτό ε, και αν απατώμε, νομίζω ότι και εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Πέλκερ και αυτό είναι ο μόνο λόγο που καθόμαστε εδώ και έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε λόγω του διαλόγου που έχουμε με τον κύριο Πόλγαρ. Δεν είναι θέμα εδώ έλλειψη εμπιστοσύνη, είναι ήδη θέμα, έλλειψη, ε, θέμα εμπιστοσύνη. Φυσικά σημείωσα όσα είπατε, αλλά δεν είναι το θέμα εδώ ότι δεν εμπιστευόμαστε ένα τον άλλον. Εμεί συζητήσαμε με τον κύριο Πόλγαρ ε, και ε, του δείξαμε κάποια εμπιστοσύνη στα πλαίσια του διαλόγου. Εμεί του εμπιστευτήκαμε. Και τώρα Νομίζω όλα υπόθηκαν. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα κατόπιν όλη αυτή τη εμπιστοσύνη. Διαφορετικά έχουμε ξοδέψει τσέπα το χρόνο μα. Totally agree with you. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Και νομίζω ότι θα του το πούμε με έναν καλό τρόπο. Βέβαια θα είμαστε κάθετοι. Ίσως κάποιος εδώ να μας ακούει προσεκτικά και να διαβιβάσει τη συζήτηση αυτή. Enttäuschen. Να το πούμε να μην μας, να μας απογοητεύσει. Μέσα Ιουνίου θα το περιμένουμε. Γιατί προ τα εκεί είχε ε, προσανατολιστεί και εκείνο για μέσα Ιουνίου. Τελειώνουμε λοιπόν, πάμε στο σημείο 14, παρουσίαση της μελέτης που είχαμε αναθέσει για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Ο κύριος Σίμων Μπροκ, που είναι ερευνητή. Είναι εδώ. Ναι, κύριε Μπροκ ευχαριστώ που θα παρουσιάσει τη μελέτη. Είμαι, ανήκω στο Παντέια, ερευνητικό κέντρο στην Ολλανδία. Θα σας παρουσιάσω την παρουσίασή μου. Καταρχάς ε, το πλαίσιο, ο στόχος της ε, μελέτης και θα δώσω κάποιες ε, πληροφορίες για το πλαίσιο αξιολόγηση που χρησιμοποίησαμε στη μελέτη. Μετά θα μπω στα πορίσματα της μελέτης και τέλος τα συμπεράσματα, συστάσεις και θα περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις για να σας απαντήσω. Ποιο είναι το πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαβίου μάθηση δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τρομέα της ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης για να προωθήσει την ε, μάθηση ε, για την κινητικότητα και τη διαβίου μάθηση. Ε, οι συστάσεις του ε, Συμβουλίου του Απριλίου του 2008 λένε ότι τα εθνικά τα εθνικά πρότυπα θα πρέπει να προσθεθούν στα ευρωπαϊκά με διαφανή τρόπο και, με την, και όπου χρειάζεται θα πρέπει να δημιουργηθούν και εθνικά πλαίσια ε, επαγγελματικών προσόντων. Το 2009 όλα τα προσόντα, διπλώματα κτλ. θα πρέπει να έχουν μια αναφορά στο, στο επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε πώς περιγράφουμε αυτά τα επαγγελματικά προσόντα στο στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να υπάρχει επίση μια διασφάλιση ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν εθνικού συντονιστέ για να υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ του εθνικού συστήματο επαγγελματικών προσόντων και του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα. Ο στόχο τη μελέτη είναι να έχουμε μια ανεξάρτητη αλόγηση για την κατάσταση, για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου, του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Ο στόχο ήταν να εξετάσουμε πώς τα κράτη-μέλη ε, αντιμετωπίζουν τις ε, προκλήσεις για την εφαρμογή αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου, ε, να έχουμε μέτρα, προσέγγιση, μια συγκεκριμένη τυπολογία μέλων, μέτρων μάλλον, και να δούμε πώς, τι δράση που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για να έχουν τα αποτελέσματα επιδιωκόμενα, για τη μεθοδολογία. Καταρχάς, συλλέγουμε δεδομένα σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, δουλειά γραφείου δηλαδή, κάναμε έξι ε, ενδελεχείς ε, μελέτες αναχώρα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία. Κάνουμε συντεύξεις με Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους και τέλος κάνουμε μία ανάλυση και συντάσσουμε και μία έκθεση. Το πλαίσιο αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε βεβαίως την τεχνική εφαρμογή των συστάσεων. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σημαντικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η μελέτη. Καταρχάς ε, το πώς σχεδιάζονται οι συστάσεις, η, τη σημασία που έχουν, τα αποτελέσματα στα οποία έχουμε καταλήξει χάρη σε αυτές. Με βάση αυτά τα τρία βήματα, σημασία, εφαρμογή και αποτελέσματα, ε, έχουμε κάποιες συστάσεις και κάποια συμπεράσματα. Αυτό είναι το πλαίσιο αξιολόγησης. Τα βασικά απορίσματα έχουμε την, ε, αυτά τα τρία στάδια που σας ε, ανέφερα και μετά θα μπω στα συμπεράσματα και στις συστάσεις. Για τα βασικά απορίσματα για τη σημασία και το σχεδιασμό των συστάσεων του πλαισίου προσόντων, θα πρέπει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να βασίζεται στη διαβίου μάθηση ε, με αυξημένη διαφάνεια για το σύστημα προσόντων και να λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές, οι γρήγορες ε, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές ε, και η παγκοσμιοποίηση ε, στον, στην αγορά εργασίας μεταξύ Ευρώπης και των χωρών. Θεωρητικά ε, πρέπει να δούμε και τη λογική παρέμβαση. Δηλαδή φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του πλαισίου αυτού είναι σαφής, έχει σαφείς στόχους, προωθεί την διαβημάθηση και την κινητικότητα των εργαζομένων και είναι σημαντικό αυτό το πλαίσιο για να, την υλοποίηση αυτών των στόχων, το πλαίσιο επαγγελματικών προσώνων. ο στόχος του είναι να προσανατολίστε στην αγορά εργασία. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια εκπαιδευτική πολιτική κατά βάση. Ε, και είναι λιγότερη σημασία του στον χώρο της εργασίας. Αν κοιτάξουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτό το EQF, ε, προωθείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκό πεδίο ε, και συνδέεται με τις ευρωπαϊκές ατζέντε, σέβεται την αρχή της επικουρικότητας παγκόσμια υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία αυτού του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Το EQF επίσης ε, συνδέεται με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εργαλεία, το ΕΚΦΕΤ, το Europass, EQUAFET, τα ευρωπαϊκά προσόντα και κατευθυντές γραμμές, ε, προσόντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, άτυπη και επίσημη διαδικασία μάθησης και όλα αυτά άλλο υποστηρίζονται και άλλο συμπληρώνονται. Αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς για να δούμε την επίπτωση αυτών των πρωτοβουλειών στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες ε, που διέπονται από την ΕΣΚΟ, ε, την ε, την οδηγία του 2005 για τα επαγγελματικά προσώτα και την αναγνώριση αυτών. Υπάρχουν δηλαδή και άλλοι τομεί. Σε σχέση με το τελευταίο αυτήν την οδηγία υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο EQF. Είναι ένα ε, σύστημα που βασίζεται στα αποτελέσματα, ενώ η οδηγία του 2005-36 έχει ένα σύστημα πέντε επιπέδων που βασίζεται πολύ στο input. Και η ευθυγράμμιση των δύο συστημάτων ε, θα ήταν καλό να γίνει. Εν συνεχεία, τα βασικά πορίσματα και την τεχνική, αν δούμε την τεχνική εφαρμογή, έχουμε, λάβαμε υπόψη μας την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Η αρχή της επικουρικότητας, όπως σας είπα, γίνεται σεβαστή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίζει το ρόλο του διευκολυντή. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά και για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη η Κομισιόν χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία και βασίζονται στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Από προηγούμενες μελέτες έχουμε εντοπίσει διάφορα, διάφορες ε, προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή και είναι η βάση α, του κεφαλαίου για την τεχνική εφαρμογή που υπάρχει στην έκθεση. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει μια προπαρασκευαστική δουλειά σε πολιτικό επίπεδο των κρατών μελών στην ανάπτυξη της πολιτικής και στις συστάσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινά μελήματα, ε, υψηλό επίπεδο συμμετοχής των φορέων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα benchmarks και οι δείκτες, ε, θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ε, και θα πρέπει να δούμε που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών ε, που τους οδηγεί ας πούμε σε αδράνεια. Όπως σας είπα, όλα αυτά περιγράφονται πολύ αναλυτικά στην έκθεση, αλλά επειδή δεν έχω αρκετό χρόνο, εγώ στέκομαι σε κάποια από τα βασικότερα πορίσματα μόνο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές αναχώρα άλλα διαφορετικά, διαφορετικά σημεία αφετηρία ό,τι αφορά την εφαρμογή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Γαλλία ξεκίνησαν τη δουλειά για αυτό το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και είχαν περιγραφεί αυτών των προσόντων και την επίπτωσή του στην μάθηση. Και ήταν εύκολο λοιπόν αυτές οι χώρες να συνεχίσουν να εργάζονται ε, επί της ε, έκθεσης ε, για το πλαίσιο. Οι νότιες χώρες όμως και οι νέες χώρες θα χρειάστηκε να αναθεωρήσουν το εκπαιδευτικό του σύστημα και να βάλουν, ε, να εισαγάγουν κάποια νέα στοιχεία στην μαθησιακή διαδικασία, κάτι που σημαίνει περισσότερη δουλειά για αυτές τις χώρες και τέλος υπήρχαν και χώρες που είχαν ε, εκπαιδευτικά συστήματα όπου κάποια μορφή προσέγγισης που να βασίζεται στα αποτελέσματα ήδη είχε εφαρμοστεί. Παρά τις ε, διαφορές ανάμεσα στις χώρες, βρήκαμε ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος για να υπάρχει διαφάνεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί μόνο χάρη σε αυτήν την αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, μπορούμε να διευκολύνουμε ε, την αγορά εργασίας. λόγω της διαφορετικής αφετηρίας των κρατών μελών υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές από χώρα σε χώρα για την διαδικασία εφαρμογής. Οι προχωρημένες χώρες έχουν ε, ξεπεράσει κάποια εμπόδια και δυσκολίες και μπορούν να βοηθήσουν άλλες χώρες για να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Οι πιο καθυστερημένες ε, χώρες ψάχνουν να δουν ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες πρακτικές και τα παραδείγματα και πώς οι πιο προχωρημένες χώρες αντιμετώπισαν τα προβλήματα. Λόγω του κοινού στόχου ή στόχων, όλες οι χώρες θέλουν ε, η εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους να γίνεται με αξιόπιστο τρόπο. Και υπάρχει μια συμβουλευτική ομάδα με συμμετοχή από όλα τα κρατημέλη και μάλιστα άλλου ενδιαφερόμενου φορεί, όπου συζητιώνται οι εμπειρίε ε, των κρατών μελών που έχουν συμμετάσχει στην ε, συγγραφή τη έκθεση και όπου ε, ετοιμάζουν κάποια σημειώματα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες Άλλο πράγμα που είναι σημαντικό είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν την πρόοδο ε, και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, για να προχωρήσει η εφαρμογή. Ένα παράδειγμα που αναφέρουμε είναι το θέμα της σύγκρισης μεταξύ των χωρών ε, για το θέμα της τετοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέλη της ε, συμβουλευτικής ομάδας επίσης, που έχουν εμπλακεί από την αρχή, ε, είναι πολύ δραστήρια, ούτω ώστε η διαδικασία να μην σταματήσει πουθενά, να συνεχιστεί και να προωθήσει τους αρχικούς στόχους. Η εφαρμογή των συστάσεων έχει πολύ σφιχτές προθεσμίες. 2010 για την έκθεση αναφοράς, 2012 για να δούμε ε, πού έχει εφαρμοστεί το, πώς έχει εφαρμοστεί το πλαίσιο ε, σε κάθε τομέα. Αυτό είναι δυνατόν, έγινε δυνατόν Μόνο χάρη στην καλή προπαρασκευαστική δουλειά όλων των κρατών μελών πριν από την σύνταξη των συστάσεων. Επίσης, αυτές οι προθεσμίες, οι σφιχτές, έδωσαν κίνητρο στα κράτη-μέλη για να δουλέψουν πιο δραστήρια, πιο ενεργά. Τα κράτη-μέλη θα είχαν ολοκληρώσει την ε, έκθεση αυτή αναφοράς ε, εμπρόθεσμα α, αν η προθεσμία ήταν τόσο κακή. Η δεύτερη, του 2010 δηλαδή. Όμως το δεύτερο, η δεύτερη προθεσμία ήταν πιο προβληματική. Πολλές χώρες δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται για τη δεύτερη φάση και οι χώρες που έχουν ολοκληρώσει την έκθεση αναφοράς δεν έχουν αναπτύξει διαδικασίες για να δείξουν πώς έχει εφαρμοστεί το EQF σε κάθε δίπλωμα, σε κάθε πιστοποιητικό. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης φάσης. Είμαστε ακόμα σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής. Και πότε θα δουν τα αποτελέσματα οι δικαιούχοι, αν δεν ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση. Αν δούμε το τρίτο τμήμα, τα αποτελέσματα, στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες επικρίσεις για την επίπτωση των, του EQF γενικά. Τις κοιτάξαμε αυτές τις επικρίσεις και πάρα είναι ενδιαφέρουσες και είναι καλό αντιστάθμισμα πολιτικής, πιστεύουμε όμως ότι το EQF δεν είναι αμφισβητήσιμο. Επίσης, μέσα σε τέσσερα χρόνια ένα τόσο μεγάλο project δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα έτσι, πλατιά. Κοιτάξαμε τρεις κατηγορίες αποτελεσμάτων, να το πω έτσι, του τι έχει γίνει τι δραστηριότητες προωθήθηκαν, ποια είναι τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, πώς συνδέονται με την αύξηση της ε, διαφάνειας και την εμπλοκή των διαφερμένων φορέων και πώς όλα αυτά αυξάνουν τη διαβίου μάθηση των εργαζομένων και την κινητικότητα των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, όλο το EQF ε, είναι ικανοποιητικό κάτι να το περισσότερο ενδιαφερομένων φορέων και προχωρεί με βάση το πρόγραμμα. Ε, δημιούργησε πολλή δουλειά, πολλές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη που συνδέεται η δουλειά αυτή με τους βασικούς στόχους των συστάσεων. Βασικό ελάττωμα. Είναι αμφισβητήσιμο αν θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η δεύτερη φάση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του EQF η αυξανόμενη διαφάνεια στη συμμετοχή των stakeholders, καλό είναι αυτό, αλλά δεν αρκεί για να υλοποιηθούν οι τελικοί στόχοι, να βελτιώσουμε δηλαδή τη διαβίου μάθηση και την κινητικότητα των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση στους βασικούς στόχους, αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατό, γιατί έχουν περάσει μόνο τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση των συστάσεων. The last Το τελευταίο τμήμα έχει να κάνει με τα συμπεράσματα. Τι βλέπουμε, ότι η εφαρμογή του QF ε, ουσιαστικά σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη δέσμευση από τους stakeholders σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και αν ε, δούμε ε, τα πρώτα αποτελέσματα την εφαρμογή του προγράμματος συμπεραίνουμε ότι η εφαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα καλό παράδειγμα μιας ε, ανοιχτής μεθόδου συντονισμού που λειτουργεί καλά. Αυτό είναι το κυρίως συμπέρασμα λοιπόν. Ε, παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, μία σειρά κρίσιμων συμπερασμάτων που πρέπει να εξαγάγουμε και αναφέρονται σε ορισμένες προκλήσεις και τεχνικά ζητήματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εφαρμογή των συστάσεων του QF για το μέλλον. ο σύνδεσμος μεταξύ του ΚΕΕΦ και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θεωρείται πολύ σαφής και πρέπει να εξηγηθεί καλύτερα πώ το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ε, θα συνεισφέρει στην επίτευξη αυτών των στόχων, περνώντα χάρη στη διαβιομάθηση. Επίσης υπάρχει έλλειψη συμμετοχής άλλων γενικών διευθύνσεων που θα έπρεπε να συμμετέχουν στην εφαρμογή του EQF, της ΓΔ για την απασχόληση και της ΓΔ Μαρκ, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερο, ένα καλύτερο προσανατολισμό προς την αγορά του EQF και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το σημείο φετηρίας και αυτέ οι διαφορές στα αρχικά στάδια επηρέασαν την πρόοδο που έγινε σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων ε, για το EQF, ε, παραδείγματο χάρη στο εθνικό, το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Επίση, υπάρχει αποκλήση μεταξύ το συστήματο 5 επίπεδου που βασίζεται στην οδηγία του 2005-36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των ε, συστήματων οκτώ επίπεδου που προκύπτουν από το EQF και συστήνουμε την ευθυγράμμιση των δύο συστημάτων. Ορισμένες τεχνικές δυσκολίες που συναντήσαμε στα κράτη-μέλη στην ε, διαδικασία Αναφορά. Αυτέ οι δυσκολίε ε, κυρίως έχουν να κάνουν με το να βρεθεί ένα σύνδεσμος ε, μεταξύ του QF ε, των συστημάτων περιορισμένη πρόοδο στο να εφαρμόζεται η προσέγγιση για την εκπαίδευση. Επίση το πώς θα συνδέσουμε τις εθνικές, τα εθνικά προσόντα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επίσης, έλλειψη διαδικασίας έγκρισης για την επίσημη και την άτυπη μάθηση, επίσης ε, διαφωνίες μεταξύ του τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης ε, και ο τρόπος ε, του πώς θα παρασχεθεί μάθηση εκτός του επίσημου τομέα και ανεπαρκής προσοχή για να ε, υποστηριχθούν τα συστήματα με διαφανείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ε, ποιότητας ε, που χρήζει για την προσέγγιση της μάθησης. Επίσης είναι δύσκολο να συμμετέχουν ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του επίσημου τομέα του εκπαιδευτικού και πιο συγκεκριμένα τους τελικούς δικαιούχους, δηλαδή τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες και κυρία χώρα είναι να συμμετέχει πλήρως η αγορά στην ε, η αγορά εργασία στην εφαρμογή σε ορισμένες χώρες ε, βρήκαμε κάτι τέτοιο, όχι σε όλες τις χώρες. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ε, τρόπο της εφαρμογής, αλλά υπάρχει και έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των εργοδοτών για την όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου επαγγελματικού Προσόντων ή για την ανάπτυξη NQF, εθνικών πλαισίων και αυτό απειλεί σοβαρά το διάλογο μεταξύ ε, του τομέα της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Ε, Πολλές χώρες επίσης ε, και συμπεριλαμβανομένων ε, όσων κατέθεσαν μία έκθεση δεν έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες να εγγυηθούν ότι η αναφορά στο κατάλληλο επίπεδο και έκθεση συμπεριληφθεί σε κάθε νέο έγγραφο σχετικά με τα προσόντα και επίσης ε, η αναφορά των εθνικών προσόντων ουσιαστικά αποτελεί ένα τεστ για το πόσο συγκρίσιμα είναι τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων ε, ένα διεθνές προσόν χωρίς ε, δράση συντονισμού θα τυθόταν στο ίδιο επίπεδο EQF από όλες τις χώρες. Αυτό πρέπει να δούμε. Ποια είναι η συνέπεια η πλήρης ε, και αξιόπιστη εφαρμογή του ΚΕΕΦ θα μπορούσε να τέθει σε κίνδυνο λόγω έλλειψης αμοιβέ εμπιστοσύνη και διαφορά ε, μεταξύ του πόσοι χώρες ε, ασχολούνται με την εφαρμογή θα μπορούσε να υποσκάψει την εμπιστοσύνη που έχουν οι χώρες στο πρόγραμμα εφαρμογής ε, των άλλων χωρών. Η αύξηση της εμπιστοσύνη εμπιστοσύνης είναι υψής της προτεραιότητας Πρέπει να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην εφαρμογή. Αυτό μπορεί να γίνει αν εφαρμόσουμε το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αναφοράς. Ουσιαστικά, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να δημιουργήσει μία όθηση ε, για να βελτιωθεί ο αντίκτυπος της όλης διαδικασίας. Αυτό το βλέπετε με την, στην ακόλουθη, επικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. Βλέπετε εδώ πώς ε, έχει τρέχουσα κατάσταση και τι συστήνουμε. Ουσιαστικά κατευθυνόμαστε προς ε, ένα προσανατολισμό ότι πρέπει να υπάρχει αυξημένη αισθήση στο δεύτερο στάδιο. Ε, έτσι λοιπόν αναμένεται ότι θα γίνουν περισσότερες συζητήσεις ε, για την εφαρμογή και ουσιαστικά θα έχουμε υψηλότερο επίπεδο δικτύπου μακροπρόθεσμα. Και φτάνω τώρα στις συστάσεις. Το Η πρώτη δέσμη συστάσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν ε, και για τα άλλα θεσμικά όργανα είναι να συνεχιστεί η εντολή του, Ευρωπαϊ... του Συμβουλευτικής για το ΚΕΦ μετά τον Απριλίο του 2013 καθώς ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η εφαρμογή του ΚΕΦ για τις μελλοντικές αγορές εργασίας και για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Επίσης, ε, στη νέα περίοδο του ΚΕΦ θα πρέπει θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική που θα απευθύνεται περισσότερο στην αγορά εργασία παρά στην εκπαίδευση και θα πρέπει να συμμετέχουν και τα ενδιαφερόμενα μέρη από την αγορά εργασίας. Αυτό δεν θα γίνει με νυχτή, αλλά πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος για το δεύτερο στάδιο, ε, ξεπερνώντας τα εμπόδια. Επίσης, μια αξιολόγηση που θα υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επόμενου μήνε, αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία άποψη που θα αξιολογεί και το παρελθόν αλλά και το μέλλον για το πώς έχει σχεδιαστεί το EQF και πώς θα εφαρμοστεί καλύτερα για να έχει καλύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Επίσης συστήνουμε να διευκρινιστεί καλύτερα πώς το EQF συνεισφέρει στους κύριου στόχους ε, της στρατηγικής του 2020 και της πολιτικής του 2020 αλλά και πρέπει να καθοριστούν και ενδιάμεσοι στόχοι. Επίσης, συστήνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αυξηθεί η συμμετοχή άλλων γενικών διευθύνσεων, όπως αναφέρα ήδη, και να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Συστήνουμε λοιπόν αυτή την περαιτέρω ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων και των πρωτοβουλειών. Και, πιο σημαντικό, θα πρέπει να γεφυρωθούν, να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της οδηγίας 2056 και του QF. Επίσης, συστήνεται στα κράτη-μέλη και στην ε, συμβουλευτική ομάδα να αυξηθεί στο δεύτερο στάδιο του referencing και επίσης ε, να οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το δεύτερο στάδιο και να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές και να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Συστήνουμε επίσης ε, να εφαρμοστεί περαιτέρω η προσέγγιση του αποτελέσματος της μάθησης ε, και να ε, συστηθούν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας για όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς. Στα κράτη-μέλη και στη διαφορετικά μέρη, σε επίπεδο κράτους μέλους, συστήνεται να αυξηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών της αγοράς εργασίας ε, για να ληφθούν περαιτέρω δεσμεύσεις, ε, να δημιουργηθεί ένα είδος οικειοποίησης ε, του EQF για τους τελικούς δικαιούχους και να προωθηθεί ένας διάλογος μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Συστήνεται να ε, ξεκινήσουν συζητήσει ε, σε επίπεδο βάση και να αυξηθεί η διαφάνεια για το πώ τα διάφορα επίπεδα συνδέονται για του τελικού δικαιούχου. Επίσης συστήνεται ε, να ε, υπάρξει ένα αποτέλεσμα μάθησης που να βασίζεται σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας για όλους τους τομείς τη εκπαίδευση και να γίνει περαιτέρω δουλειά για την επικύρωση του ανεπίσημου και του άτυπου τομέα μάθησης. Θα σταματήσω εδώ. Την έκθεση την έχετε όλοι στη διάθεσή σας. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο έγγραφο. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την έκθεση και μπροστά μας υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες σημαντικές θέματα που στη Γερμανία ενδιαφέρουν πολύ, ίσως λιγότερο σε άλλες χώρες. Ε, ας πούμε το απολυτήριο του Λυκείου δεν μπορεί να είναι ισοδύναμο με κάποιο απολυτήριο Επαγγελματική κατάρτισης πρέπει να είναι στην κατηγορία 5 το πολιτήριο, όχι 4. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλε χώρε, αλλά πάντως καλό είναι να τα δούμε όλα αυτά. Και κάποτε να τα συζητήσουμε και στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Βέβαια, μας κατακλείσατε με το κείμενο και δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα έχοντας αφομοιώσει τα πιο σημαντικά. Χρειάζεται λίγος χρόνος, εκτός και αν κάποιος μπορεί από τώρα να κάνει στοχευμένες ερωτήσεις. Δεν είναι θέμα δείγμα διαφορίας, εξηγείται ότι από το γεγονός ότι ήταν πολλά τα στοιχεία που μας δώσατε και πρέπει με την ησυχία μας να δούμε το γραπτό κείμενο, το οποίο ξεφίλησα είναι σημαντικό να το δούμε και με τους ε, φορείς ο καθένας στη χώρα του, γιατί τα προβλήματα είναι διαφορετικά σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ πολύ, θερμά σας ευχαριστώ και εσάς και τους συνεργάτες σας και πραγματικά συνιστώ να μην τη βάλετε στην άκρη την έκθεση, αλλά να την έχετε πρόχειρη και να την κοιτάτε συχνά γιατί περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες προτάσεις. Και πάμε στο τελευταίο σημείο, το οποίο το είχαμε αναβάλει από το πρωί, είναι το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών και η κατάργηση της απόφασης τάδε τάδε τάδε. Ο κύριος Φοντάνα είναι ο εισηγητής και η Ήτρε είναι επί της ουσίας ε, υπεύθυνη. Θα γνωμοδοτήσουμε εμείς. Να ακούσουμε λοιπόν τις πρωτότυπες ιδέες του κυρίου Φοντάνα για την έκθεση αυτή. Παρακαλώ, κύριε Φοντάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρα. Σα ευχαριστώ για την κατανόηση, καθώς σήμερα το πρωί δεν μπορούσα να παρευρεθώ εδώ. Και ζήτησα την αναβολή αυτού του σημείου. Θα κάνω και μία παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί δυστυχώς Ξέρετε ότι την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή μου έγινε σεισμός και σήμερα το πρωί είχαμε σεισμό και είχαμε πάρα πολλά θύματα, 15 σήμερα και νομίζω είχαμε και 6-7 νεκρούς την περασμένη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν δυστυχώς και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής πλήγει ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στην Μόδενα και έτσι λοιπόν θα αναλάβουμε κάποια δράση και με άλλους ευρωβουλευτές, Ιταλούς, γιατί Νομίζω ότι και στον πολιτιστικό τομέα θα χρειαστούμε μια βοήθεια γιατί χάσαμε ένα μεγάλο μέρος ε, των ε, θησαυρών, των καλλιτεχνικών θησαυρών αυτών των περιοχών. Είναι κάπως ιδιαίτερη η διάζωση αυτή η περιοχή. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη γνωμοδότηση. Είναι αρκετά σημαντική, γιατί αφορά τη στρατηγική για την αύξηση της ε, κάλυψης ε, της, ε, του ευρυζωνικού φάσματος στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Θέλουμε να έχουμε καθολική κάλυψη στα 30 MB ή τη σύνδεση τουλάχιστον του 50% των ε, περιμένουν με ταχύτητα άνω των 100 MB για τη διασύνδεση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση κανονισμού γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ευρώπη αν θέλει να καταστεί εκ νέου ανταγωνιστική σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να αναπτύξει και την τεχνολογία και όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της για να το κάνει και εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στο εξής. Είναι σχέδιο και μένω, γνωμοδοτησή μου, όμως ε, εγώ αυτό θα προσπαθήσω να προωθήσω, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι και ο πολιτισμό είναι μια ατμομηχανή για την ανάπτυξη τη Ευρώπη και για την οικονομική ανάπτυξη. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε η πρόταση αυτή να δίνει κάποιες ιδέες για την τεχνολογική καινοτομία και αυτή τη να έχει και ε, ουσιαστικά και μια σύνδεση με ε, τα πανεπιστήμια. Γιατί φυσικά χρειάζεται τα Ιδρύματα να έχουν τέτοιες συνδέσεις. Φυσικά η πρόταση αυτή στοχεύει στη τεχνολογική ανάπτυξη για το μέλλον. Νομίζω ότι θα γίνουν και κάποιες τροπολογίες για να προσπαθήσουμε να ευνοήσουμε και τις πιο περιφερειακές ζώνες που έχουν κάποιες δυσκολίες, όπως οι ορεινές περιοχές, παραδείγματος χάρη, οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές, περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ε, για να υπάρξει και τέτοια κάλυψη ευρυζωνική. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ είμαι ανοιχτό σε κάθε ιδέα που μπορεί να υπάρχει από τους συναδέλφους. γιατί ίσω να αναπτυχθούν καλύτερα ιδέες αν να έχουν περισσότεροι. Σε ένα μήνα περίπου θα προβούμε και στη συζήτηση 19-20 Ιουνίου και κατόπιν θα ψηφιστεί αυτή η γνωμοδότηση το Σεπτέμβριο. Εγώ ελπίζω να υπάρξει μια καλή συνεργασία, είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Νομίζω όμως ότι όλοι πάνω κάτω είμαστε υπέρ ενός τέτοιου θέματος γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και περιμένω σε αυτή την πρώτη συζήτηση τη συνεισφορά όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, την πρώτη, για την έκθεση αυτή. Ε, ζητεί κάποιος το λόγο, η Ζαμπίνε. Ορίστε. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι πολύ σημαντικά για την ε, περαιτέρω εξέλιξη των θεμάτων που μας απασχόλησαν και το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε τα απαραίτητα μέσα και στο μέλλον. Γιατί λόγω της οικονομικής κατάστασης πολλών κρατών μελών σήμερα η βελτίωση των, υποδομ... Ε, των υποδομών βραδιπορεί. Ιδιαίτερα στην Υπεθρό πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες οικονομικής προσέγγισης στην Ευρώπη, αλλά και για να αναβαθμίσουμε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Ε, το πρόγραμμα Connecting Europe, το μέσον αυτό Connecting Europe, ε, δίδει δυνατότητες, ε, προσφέρει κίνητρα και όθηση και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά εδώ της ό,τι αφορά την περαιτέρω βελτίωση των δικτύων πρέπει να δώσουμε έμφαση στην τεράστια δυναμική του προγράμματος. Το έλλειμμα των επενδύσεων είναι περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγο το ποσό. Θα χρειαστούν τα χρήματα αυτά στο καις για να ανθέξουμε και τον διεθνή ανταγωνισμό, όχι μόνο τον οικονομικό αλλά και τον πολιτιστικό. Χρειάζεται μεγαλύτερη βελτίωση. Μεγάλη δυναμική έχει και ο τομέας της εκπαίδευσης εδώ. Και η σχολική μετεκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση και η ροή πληροφοριών πέρα από το πολιτιστικό στοιχείο. δεν χρειάζεται να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή εδώ στην Επιτροπή αυτή. Ε, δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον λοιπόν να κάνουμε χωρίς τα κονδύλια αυτά και ελπίζω και από τα διορθωτικά ταμεία και από τα ταμεία ε, για την ενίσχυση της υπαίθρου να ε, μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο ίδιο πλαίσιο και το πρωί παρόμοια είπαμε αφού είναι ένα θέμα το οποίο στην καθημερινότητά μας μας επηρεάζει. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και για το σύντομο διάλογο που κάναμε, τη μικρή συζήτηση. Κύριε Φοντάν, εσείς θα συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω στην έκθεσή σας. Και ποιες είναι οι ημερομηνίε τώρα, τον Ιούνιο, στις 19 θα υποβάλλετε την έκθεση και το Σεπτέμβριο θα ψηφίσουμε την έκθεση. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι προς το συμφέρον όλων. Ε, αν σκεφτώ το πρόγραμμα e-learning, είμαστε πολύ προοδευτικοί και προχωρήσαμε. Ε, τώρα όμως χρειάζονται και τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Αλλιώς το e-learning τι να το κάνουμε χωρίς τα δίκτυα. Ευχαριστώ. Α, η Κομισιόν. Για μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Πόσο χαίρομαι που είστε μαζί μας. Ο κύριος, το όνομα, κύριος Γραμ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ χαιρόμαστε που είμαστε και εμείς εδώ, έστω και αργά που είναι. Και είμαστε στο τελευταίο σημείο. Αλλά η Κομισιόν επιμένει εδώ στις επάλξεις. Δεν έχω ε, ακούσει... Ε, να υπάρχουν ερωτήσεις από κανένα. Θέλω να ευχαριστήσω όμως τον κύριο Φοντάνα για την υποστήριξή του, για τη σύνοψη της πρότασης που αναδεικνύει την σημασία της για την τον πολιτισμό και την παιδεία, όπως είπατε κι εσείς. Το e-learning, η εκπαίδευση χρειάζονται τα ευρυζωνικά, τα ευρυζωνικά δίκτυα τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους υψηλότερες ταχύτητες, καλ, ταχύτητες, καλύτερες ε, υπηρεσίες και αντίστροφα. Η παιδεία, γενικά το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά υψηλές ταχύτητες. Όλα αυτά λοιπόν εμείς θα λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά. Ευχαριστώ που υπογραμμίσατε την σημασία που έχει αυτό για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ και εγώ την Κομισιόν. Ξέρω ότι ήρθατε και το πρωί. Ευχαριστώ πολύ που ξαναήρθατε. Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της Κομισιόν για το έργο μας. Ε, παίρνουμε μέρος της πρωινής μας κριτικής πίσω. Ευχαριστώ πολύ και η ε, υπεύθυνη συντονίστρια είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Να σας πω ότι Α, α, πρέπει να ενημερώσω για τους ε, συντονιστές που συνεδρίασαν και ε, έχετε ήδη λάβει τα αποτελέσματα της συνεδρίασης ανατέθηκε μια έκθεση, κατά τα άλλα πρόκειται για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών και για την απελευθέρωση των αποθεματικών και το ζήτημα της ηθαγένειας ή της ιδιότητας του πολίτη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα. Προσεχή συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου. Πάλι θα είναι μια ολόκληρη ημέρα, έτσι, πρωί και απόγευμα. Ευχαριστώ και καλό σας βράδυ. Ε, νομίζω τους διερμηνείς τους ευχαρίστησα ήδη. Ευχαριστούμε και εμείς.